Good afternoon, colleagues. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ που ήρθατε καιρός. Ξέρω ότι είναι πέμπτη απόγευμα, γι' αυτό και περίμενα λίγο, αλλά έχουμε ένα πολύ σημαντικό σημείο στην ημερήσια διάταξη και χαίρομαι που καταφέρατε και ήρθατε. Το θέμα λοιπόν είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Julian King, αρμόδιο για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι που ήρθε. Είχαμε το αναβάλει ήδη μια φορά και χαίρομαι που επιτέλους καταφέραμε να οργανώσουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ θερμά και τον Επίτροπο αλλά και εσάς για την υπομονή σας και επίσης σας ευχαριστώ για όσοι συμμετείχαν στην προπαρασκευαστική συνεδρίαση για να ετοιμάσουμε τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων. Και ευχαριστώ και την Μπάρμπαρα που προέδρευσε σε εκείνη την προπαρασκευαστική συνάντηση. Ο διορισμός του Επιτρόπου Κίνγκ ως αρμοδίου Επιτρόπου για την Ασφάλεια της Ένωσης και σε συνδυασμό με την κατεπίγουσα ανάγκη της βελτίωσης της ασφάλειας στην Ευρώπη μας οδήγησε να συστήσουμε στην Επιτροπή Πολιτικής πολιτικών ελευθεριών ένα πιο διαρθρωμένο διάλογο για την ασφάλεια μεταξύ της Επιτροπής μας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Προεδρίας του Συμβουλίου και εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη. Και είπαμε ότι τέτοιος διαρθρωμένος διάλογος θα πρέπει να λαμβάνει χώρα τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, ώστε να έχουμε το, το χρόνο για μια ευρυθέστερη, σφαιρικότερη και πιο εμπαριστατωμένη συζήτηση για ειδικά θέματα του τομέα ασφάλειας ο πρώτος ε, διάλογος για την ασφάλεια με τον Επίτροπο King θα περιστραφεί γύρω από την ε, εφαρμογή και χρήση των ε, υφισταμένων εργαλείων για την ανταλλαγή πληροφοριών στα θέματα ασφάλειας. Νομίζω ότι έχει νόημα μια πιο διεξοδική συζήτηση για τα θέματα αυτά. Τον ευχαριστώ και για τα έγγραφα που μας έστειλε για να προετοιμάσουμε τη σημερινή μας ακρόαση και Ευχαριστώ, επαναλαμβάνω και όσοι συμμετείχαν στην ε, ε, προπαρασκευαστική συνεδρίαση της 6ης Μαρτίου με ε, εθνικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας και εφαρμογής του νόμου. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον Επίτροπο για να μας κάνει μια εισαγωγή. Ίσως θα μιλήσει και για τις επιθέσεις στο Λονδίνο και την επέτειο που είχαμε χθε για τις τρομοκρατικές επιθέσεις των Βρυξελών και μετά να μας παρουσιάσει το θέμα του. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας καταρχήν. Και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να πω πρώτα δύο λόγια για τα χθεσινά συμβάντα. Πριν περάσω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Φαντάζομαι ότι μιλώ στο όνομα όλων Λέγοντα ότι η επίθεση χθε σε πεζούς που περνούσαν από μία γέφυρα, την γέφυρα Westminster στο Λονδίνο και η επίθεση και στο Κοινοβούλιο του Λονδίνου μας άφησε συγκλονισμένους, αναβδούς και φυσικά ε, η σκέψη μας ε, πηγαίνει κυρίως στα θύματα. Δεν νομίζω ότι ήταν τελείως τυχαίο που η επίθεση αυτή έλαβε χώρα κατά την πρώτη επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων στις Βρυξέλλες. Όταν εδώ, στην πρωτεύουσα του Βελγίου, ε, τιμούσαμε τη μνήμη των 32 θυμάτων ε, και των πολλών ε, τραυματιών που άλλαξε η ζωή τους μετά την επίθεση των Βρυξελών. Η μεθοδολογία μάλιστα του αυτούργου της επίθεσης του Λονδίνου ακολουθεί ένα τρόπο συμπεριφορά που δεν ήταν καινούριο. Έγινε πέρυσι στην Νίκαια, στην Εθνική Ορτή τη Γαλλία, αλλά και στο Βερολίνο λίγο πριν τα Χριστούγεννα. μετατρέποντα ένα όχημα, ένα καθημερινό αντικείμενο, σε όπλο κατά του ευκολότερου στόχου των απλών ανθρώπων που ζουν την καθημερινότητά τους και που δεν δημιουργούν απειλή για κανένα στον κόσμο. Ε, μάλιστα, είδαμε από την τελευταία επίθεση ότι εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή η τρομοκρατική απειλή παντού στην Ευρώπη. Η επίθεση αυτή ολοκληρώθηκε στον περίβολο του ε, Βρετανικού Κοινοβουλίου και συνιστά μια απειλή στην ίδια τη δημοκρατία. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που συμμεριζόμαστε όλοι, έτσι αντιλαμβανόμαστε όλη αυτή την επίθεση. Και η, η αυτούργη της επίθεσης αυτής ε, έπληξαν την καθημερινότητά μας, τις αξίες μας, ε, την εργασία μας. Δεν θα τους αφήσουμε όμως να κερδίσουν, δεν θα πτωηθούμε. Και όπως και η Γαλλία αποφάσισε πέρυσι να οργανώσει το πρωτάθλημα του 2016 το ποδοσφαιρικό, παρά της, ε, την επίθεση στην Νίκαια, και οι γερμανικές αρχές αποφάσισαν στο Δεκέμβριο να κρατήσουν ανοιχτές τις χριστουγεννιάτικες αγορές παρά την τρομοκρατική επίθεση, με ενισχυμένα βέβαια μέτρα ασφάλειας, αλλά δεν το ήθηκαν. Και ποτέ δεν θα αποκαταστήσουμε ασφάλεια 100%. Ούτε ποτέ θα εκμηδενήσουμε τον κίνδυνο της επίθεσης. Αλλά μπορούμε και οφείλουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να καθιστούμε όλο και δυσκολότερες τις ε, επιθέσεις αυτές, την ενέργεια τέτοιων ενεργειών. Και πιστεύω ότι πραγματικά σημειώνουμε πρόοδο στην προσπάθειά μας, σε αυτή την κοινή, τη συλλογική προσπάθεια που κάνουμε να περιορίσουμε τις δυνατότητες ε, των τρομοκρατών και άλλων να μας βλάψουν. Και ε, συνεργαζόμαστε για να γίνουμε όλο και πιο ανθεκτικοί σε τέτοια πλήγματα. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, γιατί αυτό που συζητούμε σήμερα ακριβώς είναι μια πτυχή αυτού του έργου που συνεχώς πραγματοποιείται. Θα περάσω τώρα στο θέμα που είναι το αντικείμενο της ε, σημερινής μας ημερήσιας διάταξης. Είπαμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη συζήτηση για να μιλήσουμε για διάφορα εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών στα πλαίσια της προσπάθειας ενίσχυσης ε, της κοινή μας ασφάλειας. Και χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω αυτά τα εργαλεία. Μάλιστα σας έστειλα και κάποια προπαρασκευαστικά έγγραφα, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Και από ό,τι κατάλαβα είχατε και μια πολύ παραγωγική ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων με εθνικού εμπειρογνώμονε. Οι απειλέ γίνονται όλο και πιο περίπλοκε και πολυσύθετε. Γι' αυτό και η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών γίνονται πιο σημαντικέ από ποτέ για να ενισχύσουμε πραγματικά την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Μόνο από κοινού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις απειλές και τις τρομοκρατίες αλλά και το οργανωμένο εγκλήματος και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Όπως είπα και προηγουμένως, ε, πιστεύω ακράδαντα ότι το πρώτο βήμα είναι να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την υπάρχουσα νομοθεσία και τις υφιστάμενες ε, πρωτοβουλίες για να προωθήσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των ε, φορέων και παραγόντων στον τομέα της ασφάλειας. Γι' αυτό η Κομισιόν ζητά συνεχώ από τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν πλήρω το δυναμικό των υπαρχόντων συστημάτων ανταλλαγή πληροφοριών και συνδράμουμε τα κράτη-μέλη με χρηματοδότηση, με εμπειρογνωμοσύνη και με κοινοποίηση των βέλτιστων πρακτικών. Μάλιστα, την τελευταία διετία προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση και τον Απρίλιο του 2016 συστήσαμε μια στρατηγική για τα συστήματα πληροφοριών και ασφάλεια των συνόρων με την ανάλυση υπαρχών των συστημάτων πληροφοριών και εντοπίζοντας τις αδυναμίες και τα κενά τους προκειμένου να προτείνουμε δράσεις για να τα αντιμετωπίσουμε. Η καλύτερη εφαρμογή και χρήση των συστημάτων πληροφόρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ε, πρόκλησης ε, να εξασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα και στιβαρά συστήματα πληροφοριών. Και μάλιστα και το Φεβρουάριο είχαμε σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια. Για όσου όμω αποσίαζαν από την περίπτωση εκείνη, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη ανακεφαλαίωση. Πώ έχει η κατάσταση για τα υπάρχοντα συστήματα, τα υφιστάμενα συστήματα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το σύστημα πληροφοριών Schengen. Αυτή είναι η ευρέω χρήση ε, βάση πληροφοριών στην Ευρώπη και πραγματικά είναι πολύ ε, επιτυχής η πρωτοβουλία αυτή και χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από τα κράτη-μέλη. Χρόνο με το χρόνο αυξάνεται η χρήση. Ε, μάλιστα το 2016 είχαν περίπου 4 ε, δισεκατομμύρια επισκέψεις δηλαδή σε δεδομένα. Δηλαδή αύξηση κατά 40% σε σχέση με τη χρήση του 2015. Και μάλιστα τα hits ήταν από 50.000 ε, το 2015, 200.000 το 2016 οι αναζητήσεις. Και βέβαια σίγουρα υπάρχει δυνατότητα για τεχνικές και επιχειρησιακές ε, βελτιώσεις για να γίνει το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν πιο αποτελεσματικό. Και γι' αυτό και καταθέσαμε μια σειρά νομοθετικών προτάσεων, τις οποίες θα σας εξηγήσω εντός ολίγου. Πάντως, ε, η οργανισμός, η Γιουλισσάς, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις τεχνικές βελτιώσεις ε, του ΣΥΣ και κυρίως ένα σύστημα ε, αυτοματοποιημένης ε, λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων του ΑΦΙΣ, ώστε να μπορούν τα όργανα επιβολής νόμου να αναζητήσουν υλικό δακτυλικών αποτυπωμάτων στο σύστημα. Έτσι γίνεται πιο αξιόπιστη εξακρίβωση των στοιχείων για να εμποδίσουμε ως ταξιδεύουμε πλαστές ταυτότητες. Και μάλιστα ε, μέχρι τα τέλη του χρόνου θα έχουμε τη συμμετοχή 6 πλέον χωρών μελών. Και μάλιστα θέλουμε να ε, έχουμε εξτρατεί συνειδητοποίηση στα κράτη-μέλη και αυτό βοήθησε στην αύξηση του αριθμού των ελέγχων και την αυξημένη χρήση από τις εθνικές υπηρεσίες του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν και μάλιστα με πιο μακροπρόθεσμη προοπτική είχαμε αύξηση κατά 800% του αριθμού των συγκεκριμένων προειδοποιήσεων για έλεγχο από τις εθνικές ε, υπηρεσίες ασφαλείας τα τελευταία χρόνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις ΠΡΙΜ, όπως ξέρετε, οι αποφάσεις ΠΡΙΜ είναι σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας. Ξεκίνησε το 2008, ε, προβλέποντας ανταλλαγή στοιχείων για το DNA, ε, της άδειας κυκλοφορίας ε, και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Ο Αύγουστος του 2011 ήταν η καταληκτική προθεσμία ε, για την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη, αλλά πέντε χώρες δεν έχουν ακόμη τηρήσει τις αποφάσεις πριν. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε στην Επιτροπή το περασμένο Σεπτέμβριο διαδικασίες σε παραβάση. Έχουμε λάβει τις απαντήσεις των πέντε χωρών μελών και τις επεξεργαζόμαστε πριν περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Εκ παραλλήλου, βοηθούμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο τις αποφάσεις Πριν με χρηματοδότηση και ανταλλαγή των πρακτικών. Επίσης, Σουηδική πρωτοβουλία. Όπως ξέρετε, προτείνει ένα κοινό νομικό πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Ήταν καλή η πρόοδο στην εφαρμογή, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν αυτή την πρωτοβουλία της Σουηδία στα κράτη-μέλη ε, για να γίνει μια αξιολόγηση συμμόρφωσης ε, είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο για να δημιουργήσουμε μια γενική εικόνα της κατάστασης και να δούμε ποια θα είναι τα βήματα για να εξασφαλίσουμε πλήρη εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Επίσης, η, συμβουλία, η απόφαση 671 του Συμβουλίου για την ανταλλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά τρομοκρατικές ενέργειες με παροχή πληροφοριών στην Ευρωπόλα, Eurojust και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη ε, υπό τον όρο ότι δεν διακυβεύουν ε, τρέχουσες έρευνες. Και αυτές οι υποχρεώσεις ενισχύθηκαν από την υιοθέτηση και τις οδηγίες ε, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και θα ήθελα ευκαιρία να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως τη δική σας Επιτροπή για το έργο σας και την συνεισφορά σας στο θέμα αυτό, που θα συμβάλλει περαιτέρω στην ενίσχυση της ασφάλειας. Πέμπτο θέμα, το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις, VIS. Επίσης, θέτει κάποιες ασφαλιστικέ δικλείδε. Από το Σεπτέμβριο του 2013 οι αρχέ επιβολή του νόμου είχαν πρόσβαση σε αυτή τη, βάση, αυτή τη βάση δεδομένων του ΒΙΣ με βάση μια συγκεκριμένη απόφαση για την εφαρμογή του νόμου. Και μάλιστα μια αξιολόγηση που πραγματοποιήσαμε κατέδειξε ότι η πρόσβαση στο ΒΙΣ ε, για τη, θε, λόγους νόμου είναι κατακαιρματισμένη προς το παρόν. Σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς, Είχαμε σημαντική πρόοδο την τελευταία διετία σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με την, Euro, με την Ευρωπόλ και την Eurojust. Για παράδειγμα, οι ξένοι μαχητές και τα στοιχεία για αυτούς προς την Ευρωπόλ με στόχο να μπουν στο σύστημα της Ευρωπόλ έχει διπλασιαστεί από το Σεπτέμβριο του 2015. Ήταν 7.800 οι είσοδοι νέων ονομάτων με Ευρωπαίους υπηκόους και υπηκόους τρίτων χωρών. Κάτι που αυξάνει την εμπιστοσύνη στα συστήματα της Ευρωπόλ. Βέβαια, θα, πρέπει να, γίνει, να λαφθεί υπόψη και η επιχειρησιακή τους αξία. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα, το, δελ, το Μητρό Ονομάτων Επιβατών. Έχει συμφωνηθεί από όλους, αλλά δεν εφαρμόζεται ακόμη πλήρως από όλους. Έχουν μέχρι το Μάιο του 2018 τα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν τη σχετική οδηγία για το PNR και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πέρυσι τον Νοέμβριο ένα σχέδιο εφαρμογή με κατευθυντήριε γραμμέ και τι βέλτιστε πρακτικέ. Και μάλιστα οργανώσαμε σεμινάρια, ειδικέ συνεδριάσει και θα παράσχουμε χρηματοδότηση καθώ και μια ειδική πλατφόρμα για του ε, ειδικού. Επίσης θα υιοθετήσουμε και μια εκτελεστική απόφαση για τα φόρμα των δεδομένων και τα πρωτόκολλα Διαβίβασή του που θα πρέπει να τηρούν οι αεροπορικέ εταιρείε όταν ε, μεταβιβάζουν στοιχεία PNR στι αρχές των κρατών μελών. Τώρα να περάσω στις νομοθετικές πρωτοβουλίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις οποίες παρουσιάζουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα κενά που διαπιστώσαμε στη στρατηγική του 2016 η Επιτροπή παρουσίασε τρεις προτάσεις το Δεκέμβριο για να βελτιώσουμε τη χρήση του SIS, του Συστήματος Πληροφοριών Σέγγεν και αυτά θα πρέπει να συνεχίσουν να επιτρέπουν αποτελεσματική ανταλλαγή μεταξύ κρατών μελών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο διασυνοριακό έγκλημα. Για πρώτη φορά προτείνουμε να είναι υποχρεωτικό τα κράτη-μέλη να εκδίδουν alert στο SIS για άτομα τα οποία σχετίζονται με τρομοκρατικά ε, εγκλήματα. Επίσης, ε, θέλουμε να έχουμε και απαγόρευση εισόδου για υπηκόους τρίτων χωρών που βρίσκονται στο SIS ε, για να ενισχύσουμε την εφαρμογή αυτών των απαγορεύσεων. Θέλουμε να ενισχύσουμε επίσης την προστασία δεδομένων με επιπλέον δικλείδες ασφαλείους βάσει των θεωρημένων κανόνων για την προστασία δεδομένων. Αυτά τώρα είναι προς το Συμβούλιο για συζήτηση και φυσικά προσβλέπω και στη στενή συνεργασία με τους εισηγητές για να προωθήσουμε όλα αυτά τα θέματα μαζί σας. Άλλες προτάσεις που έχουμε επιτάπητος αφορούν τη μεταρρύθμιση της βάσης δεδομένων ασύλου, τη Eurodac, για να βελτιώσουμε περαιτέρω τις ε, λειτουργίες τους όσον αφορά την ε, παράτυπη μετανάστευση και τις επιστροφές και την επέκταση του ε, συστήματος ποινικού μητρώου για να το επεκτείνουμε και σε επικόστριο των χωρών. Θα προ είναι η Επιτροπή μια τροποποιημένη πρόταση τον Ιούνιο. Να σας πω και δύο λόγια για την πρόταση για ένα σύστημα εισόδου-εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα καταγράφει ε, ποιοι υπήκοοι των χωρών περνούν τα εξωτερικά σύνορα Σέγγεν. Πιστεύουμε ότι θα βελτιώσει την ασφάλεια και ε, θα λέει φυσικά και στις αρχές των κρατών μελών ποιοι ε, εισέρχονται, ταξιδεύουν και αποχωρούν από το χώρο Σέγγεν. Και για να καταπολεμήσουμε και το σοβαρό έγκλημα θα υποστηρίζουμε την εξακρίβωση των υπόπτων και φυσικά υποστήριξη και προς τα θύματα. Χαίρομαι για την πρόοδο που επετεύθη από τον εισηγητή, τον κύριο Ντίας Τεμέρα και την Επιτροπή σας για τα θέματα αυτά και περιμένουμε φυσικά να ε, ολοκληρωθούν όλες αυτές οι εργασίες. Τέλος, να σας πω και δύο λόγια για την πρότασή μας για ένα ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και έγκρισης, το ETIAS θα μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε την ασφάλεια και την, ε, τους κινδύνους της παράτυπης ε, για τους υπηκόους τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από τη θεώρηση διαβατηρίου πριν ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπιστώνοντας ποιοι είναι πιθανοί υποπτοί και απαγορεύοντας τους ε, την είσοδο, ε, θα αυξήσουμε την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και όπως είπαμε και στην κοινή δήλωση, η πρόταση είναι νομοθετική προτεραιότητα και λογικά θα πρέπει να εγκριθεί πριν από το τέλος του έτους και με τα χαράς ε, να υποστηρίξω και την εισηγήτρια, την κυρία Γκάλ, ε, σε οποιαδήποτε προσπάθεια χρειάζεται προκειμένου να προωθεί το ζήτημα. Είπαν κάποιοι ότι το έργο για το ΕΤΙΑΣ εξαρτάται και από την πρόοδο που θα επιτευχθεί στις συζητήσεις για τη διαλειτουργικότητα. Αλλά θα ήθελα να σας πω σήμερα το απόγευμα ότι εγώ δεν είμαι βέβαιος κατά πόσον ε, ισχύει κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση ΕΤΙΑΣ το Νοέμβριο του 2016 για να αντιμετωπίσει ένα πολύ σημαντικό κενό πληροφοριών για τους ταξιδιώτες που απαλλάσσονται από τη θεώρηση διαβατηρίων και αυτό το κενό απαιτεί συγκεκριμένη δράση για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα το ΕΤΙΑΣ είναι αυτόνομο εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει να πληρωθεί αυτό το κενό, ανεξάρτητα από το τι κάνουμε εκ παραλλήλου σε θέματα διαλειτουργικότητας. Λόγω του γεγονότος ότι πρέπει να δράσουμε κατεπηγόντως για το ΕΤΙΑΣ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε εξαίρεση και δεν υπέβαλε εξολόγηση επιπτώσεων. Ξέρω ότι κάποιοι από εσά είχατε ερωτηματικά επ' αυτού, αλλά βασίσαμε την πρότασή μας σε μια πλήρη μελέτη σκοπιμότητας, η οποία δημοσιεύτηκε από κοινού με την πρόταση και βεβαίως ακριβώς λόγω του κατεπήγοντος ε, χαρακτήρα ε, αυτού του, της πλήρωσης αυτού του κενού όλα τα θεσμικά όργανα συμφώνησαν να γίνει προτεραιότητα του ΕΤΙΑΣ ε, στην κοινή δήλωση. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνουμε για τη διαλειτουργικότητα δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να καθυστερήσει σημαντική δουλειά για πράγματα τα οποία συζητώνται αυτή τη στιγμή από τους συνομοθέτες, μεταξύ των οποίων και το ΕΤΙΑΣ, το σύστημα εισόδου-εξόδου και την πρόταση για την ενίσχυση του SIS. Δεν επηρεάζει ούτε καθυστερεί τις εργασίες για αυτά τα συστήματα πληροφοριών, τα οποία ούτως ή άλλως χρειαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να τα χρειαζόμαστε, ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίσουμε στη συνέχεια από κοινού να κάνουμε για τα θέματα διαλειτουργικότητας. Ε, γεγονός που με φέρνει και στο τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να θίξω. Τα όσα κάνουμε για τη διαλειτουργικότητα, για να μπορέσουμε να συνδέσουμε καλύτερα πληροφορίες μεταξύ των διαφόρων πληροφοριακών μας συστημάτων. Την τελευταία φορά που ήμουν εδώ στην Επιτροπή σας, στα τέλη Ιανουαρίου, ε, με πολύ χαρά συζήτησα μαζί σας ε, ό,τι βρήκαμε για την ομάδα υψηλού επίπεδου για τα συστήματα ε, πληροφορικής και τη διαλειτουργικότητα. Η ομάδα που συστήθηκε για να εξετάσει τις διάφορες εναλλακτικές επιλογές για τη διαλειτουργικότητα συνεχίζει τις εργασίες της και θα υποβάλουμε τελική έκθεση στις αρχές Μαΐου με ό,τι έχουμε διαπιστώσει και τις σχετικές μας συστάσεις. Στη συνέχεια και βάσει και τη στρατηγική μας του Απριλίου του 2016 η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει συγκεκριμένε ιδέες και σε εσά στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στα μέσα Μαΐου, τα οποία θα αποτελέσουν και βάση για συζήτηση μαζί σας για το τι μελιγενέστε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, συγγνώμη που μακρηγόρησα και είμαι στη διάθεσή σας για τη συζήτηση σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. που έχουμε αυτό το διάλογο μαζί σας και Χαίρομαι που προσήλθαν τόσοι πολλοί ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής μας σήμερα σε αυτή την συνεδρίασή Μα Νομίζω ότι ε, αναφερθήκατε σε ζητήματα που μας απασχολούν και μας ανησυχούν όλους. Είναι μεγάλος ο κατάλογος ομιλητών, αλλά έχουμε χρόνο. Πρώτα θα ακούσουμε τους συντονιστές. Ο κύριος Ρομπέτο Μετσόλα έχει το λόγο. Κυρία, ευχαριστώ Σα ευχαριστώ για αυτή την πολύ ολοκληρωμένη παρουσίαση για το τι μελή γενέστε και τις δράσεις που πρόκειται να λάβει η Κομισιόν στον τομέα σα. Καθώς οι χθεσινές ε, επιθέσεις έγιναν την πρώτη επέτειο των επιθέσεων στις Βρυξέλλες, πρέπει πραγματικά να ε, είμαστε διαρκώς σε εγρήγορση λόγω του υψηλού κινδύνου τρομοκρατίας που αντιμετωπίζουμε στις χώρες μας και γι' αυτό ε, συνεχίζουμε και ως ε, ομάδα να καλούμε την Επιτροπή να αναλάβει δράσεις προκειμένου να παραμείνει η ασφάλεια σε υψηλότερο επίπεδο. Έχω κάποια ερωτήματα για να μπούμε σε λίγο περισσότερε λεπτομέρειε σε σχέση με αυτά που μα είπατε. Όσον, αφορά το πιλωτικό πρόγραμμα για τα δακτυλικά αποτυπώματα, αναφερθήκατε σε έξι κράτη-μέλη. Μπορείτε να μα πείτε λίγα περισσότερα πράγματα όσον αφορά μια ενδεχόμενη επέκταση του πιλωτικού αυτού προγράμματος και σε άλλες ε, χώρες ή οτιδήποτε μας πείτε ε, επί του θέματος αυτού και για την πρόοδο που σημειώνεται θα είναι χρήσιμο. Ε, για το Νομίζω ότι είναι πραγματικά κρίμα που δέκα χρόνια μετά την έγκρισή του τόσα πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην πλήρη εφαρμογή του. Είναι ένα εργαλείο που θεωρήσαμε τότε ότι ε, θα ήταν κάτι που θα βοηθούσε στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών και αυτό ε, ε, ήταν κάτι που το επιδιώκαμε ε, στις προσπάθειές μας στα κράτη-μέλη. Για το αίτιας ε, χαίρομαι που αναφερθήκατε στο ζήτημα της μελέτης επιπτώσεων. Χθες είχαμε μια πολύ μακρά συζήτηση με, εδώ στην Επιτροπή για το αν η μελέτη επιπτώσεων και σκοπιμότητας αρκεί. Εμείς θεωρούμε ότι ε, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα ε, αυτή η κάλυψη του κενού που καλείται να, ε, υλοποιήσει, να υλοποιηθεί με το αίτιας. Παρόλα όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες για το αν αυτή η πρόταση μπορεί να προχωρήσει χωρίς μελέτη Παρ' όλα αυτά ε, προσβλέπουμε στα πορίσματα της ειδική ε, ομάδας της Task Force τον Μάιο και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δούμε πιο στενά τις ε, συγκεκριμένες συστάσεις που θα γίνουν. Κυρία Ζήπελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κίνγκ που βρίσκεστε εδώ. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, μπερδεύομαι και λίγο ενοχλούμε από τα συνεχή, τις συνεχείς εκκλήσεις ότι πρέπει να κλείσουμε τα κενά και τα και τα λοιπά ε, και ότι γι' αυτό και την επιτακτική ανάγκη και γι' αυτό δεν υπήρξε μελέτη επιπτώσεων. Ε, θυμάμαι ότι στις επιθέσεις των Βρυξελών ένα από τα προβλήματα που είχαμε αντιμετωπίσει ε, όσον αφορά την ε, εξέβρεση πληροφοριών για κάποιους τουλάχιστον από τους δράστες ήταν το γεγονός ότι δεν είχε χρησιμοποιηθεί επαρκώς το SIS. Είπατε ότι η απόφαση πριν έπρεπε να είχε ε, εφαρμοστεί από το 2011, ενώ υπάρχουν ακόμα κράτη-μέλη που δεν το κάνουν και η διαδικασία που παραβάσει ξεκίνησε μόλις το 2016. Επίσης είχαμε κάνει μια συζήτηση για την συνοριοφυλακή και την ακτοφυλακή, όπου μας βιάσατε να λάβουμε την απόφαση και τώρα μαθαίνουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις τους. Άρα γιατί βιαζόμαστε κάθε φορά, αν σε τελική ανάλυση βλέπουμε ότι όλες αυτές οι αποφάσεις δεν εφαρμόζονται. Το ίδιο ισχύει και για το Eurodac. Τώρα θα προετοιμάσουμε μια ε, απόφαση για τη συλλογή ακόμα περισσότερων πληροφοριών, ενώ εγώ προσωπικά δεν έχω δει ακόμα την ε, μελέτη επιπτώσεων ε, για το κατά πόσο τελικά θα ε, είναι χρήσιμη η λήψη δεκτυλικών αποτυπωμάτων από παιδιά 6 ετών. Δεν ξέρω σε ποιον βαθμό ε, θα είναι χρήσιμο, καθώς τα δακτυλικά αποτελέσματα από τους ετούντε άσυλων δεν καταχωρίζονται πάντοτε στο, στο Έχουμε διάφορα κενά πληροφοριών, τα οποία τα δημιουργούν τα ίδια τα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά, εμείς ζητούμε όλο και περισσότερες λεπτομέρειες, όλο και περισσότερες πληροφορίες. Πραγματικά, ανυπομονώ πέντε χρόνια από σήμερα να δω τι πρόοδο θα έχει σημειωθεί ε, σε σχέση με το αίτια ή αν ε, ξαναέρθουμε εδώ να, διαμορφω... να διαμαρτυρηθούμε για τα κενά πληροφοριών και για την έλλειψη ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Εν πάση περιπτώσει, επί της αρχής, μιλώντας για την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα του συστήματος, δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, λέμε ότι θέλουμε περισσότερα δεδομένα, από την άλλη όμως έχουμε και, τις, ε, και, την, ε, και το σημείο καμπής που μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε υπερβολικά πολλά δεδομένα και στη συνέχεια ε, χρειάζεται να έρθουν σε επαφή άνθρωποι για, το, για, για τα ονόματα των επιβατών. Και ε, μας είχαν πει ε, σε μια ακρόαση που είχε διοργανωθεί εδώ ότι ε, χρειάζονται εκατομμύρια φίλτρα προκειμένου να μπορέσει κανείς να ανοιχνεύσει εκείνες τις πληροφορίες που θα βοηθήσουν τις αρχές στο να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Παρ' όλα αυτά όμως και παρόλα, παρόλα αυτά εμείς έχουμε δημιουργήσει και άλλες υποχρεώσεις συλλογής πληροφοριών. Ωστόσο, αν το κάνουμε αυτό. Πώς μπορεί η Κομισιόν να εξασφαλίσει τόσο την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων αλλά και τις ε, διαδικαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, τις δικαστικές ε, ασφαλιστικές δικλείδες, την ε, νομική, τα ένδικα μέσα ή το τεκμήριο της αθεότητας. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πρόταση να δημιουργηθεί μια κοινή βάση δεδομένων που θα καταχωρίζονται όλα τα δεδομένα Είχαμε και χθε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν και κατά πόσο ε, είναι χρήσιμο να συλλέγονται όλα τα ποινικά δεδομένα, τα δεδομένα για την υγεία, ε, παρά το γεγονός ότι ε, αντίστοιχες διαδικασίες ακολουθούν η Ιντερπολ και η Ευρωπόλ. Τέλος, μιλώντας για τη διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία ενός αποθέματος δεδομένων, αναμένουμε, μπορούμε να αναμένουμε κάποια νομοθετική πρόταση ε, όταν πια δημοσιευτεί και η τελική έκθεση της ομάδας υψηλού επίπεδου και μπορείτε να μας ε, υποσχεθείτε ότι εν ώψη μιας τέτοιας πρότασης θα υπάρξει και μια πραγματική διοργανική ε, διαβούλευση και ότι θα συνοδεύεται μια τέτοια νομοθετική πρόταση και από μια πραγματική μελέτη επιπτώσεων. Ευχαριστώ. Η κυρία Στήμας χρειάστηκε να φύγει, αλλά φαντάζομαι ότι θα επανέλθει. Κυρία Φράουντ Νάταλη. Η κυρία Γκρισπέκ, Ευχαριστώ Κλοντ, ευχαριστώ κύριε πίτροπε. Αυτή η πρώτη συζήτηση για τον πρώτο διάλογο για την εσωτερική ασφάλεια και η σημερινή ανταλλαγή απόψεων είναι ζωτική σημασίας μετά από ε, αυτά τα διπλή ε, συμβολική χθεσινή ημέρα, από τη μια την επέτειο των τρομικρονικών επιθέσεων στις Βρυξέλλες και από την άλλη ε, τα ε, αποτρόπαια χθεσινά γεγονότα στο Λονδίνο. Ε, από ό,τι βλέπετε κύριε Επίτροπε είναι πολύ σημαντικό το χαρτοφυλάκιό σας και πόσο σημαντικό επίσης οι Ευρωπαίοι πολίτες να λάβουν και μία απάντηση από πλευράς ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σε θέματα ασφαλείας και κυρίως σε ποιοτικά στοιχεία όσον αφορά την Ευρώπη. Ελπίζω ότι από εδώ και πέρα μέχρι την επόμενη διετία, γιατί η θητεία σας μέχρι τότε θα διαρκέσει ε, και ε, θα τελειώσει φυσικά και η θητεία των Ευρωβουλευτών. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να ε, παραδώσουμε κάποια πράγματα, να έχουμε κάποια απτά αποτελέσματα κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, την αναφέρετε στην εισαγωγή σας ε, και όλοι το γνωρίζουν σήμερα. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι ένας τομέας στον οποίο ακόμα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης, ε, διότι πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος είναι ακόμα γεμάτος κενά, ε, Εμβαλωματικό, υπάρχουν ε, προβλήματα ποιότητα για την ανταλλαγή δεδομένων και προβλήματα ανταλλαγή πληροφοριών, πρόσβασης ε, δεδομένα επιτόπου και από την άλλη είναι και τμηματική γιατί δεν δίνει λύσεις σε κάποια πράγματα. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχουμε διαπιστώσει. Χρειαζόμαστε περαιτέρω κονδύλια για την εσωτερική ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, ε, ένα ενιαίο ε, πεδίο ε, interface αναζήτησης. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τι κάνουμε όμω, κύριε Επίτροπε για να προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα. Δεύτερον, όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων και κάποιων ε, δράσεων και τη νομοθεσία, ε, στην ακρόασή σας είχατε πει ότι θα πρέπει να γίνει μια συνολική αξιολόγηση. Ε, θα γίνει αυτή η συζήτηση προσεχώ στις 3 Απριλίου και ελπίζω και από την ομάδα σας, με αυτό σας ζητώμε, να δώσετε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, να υπάρξουν ε, ε, δράσεις μετά από αυτή την αξιολόγηση για να μπορέσουμε να τα μεταφράσουμε σε απαντήσεις και να προχωρήσουμε. Τρίτο, όσον αφορά την, ε, το κυβερνοέγκλημα, θυμάμαι στην ακρόασή σας, ε, μου άρεσε ιδιαίτερα ο όρος που χρησιμοποιήσετε ε, στα γαλλικά για την προσαρμοστικότητα σε επίπεδα, σε θέματα κυβερνοασφάλειας. θεωρήσαμε ότι αυτή θα πρέπει να είναι μια πραγματική πολιτική δράση και να ρωτήσω λοιπόν τι συγκεκριμένο έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πίσω από αυτό τον όρο της κυβερνοπροσαρμοστικότητας ε, και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, εσείς πώς θα προσαρμόσετε τις δράσεις σας. Και τέλος, ε, κάτι πολύ επίκαιρο, ε, πριν από 48 ώρες, οι Ηνωμένε Πολιτείε επέβαλαν νέους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ε, ταμπλέτας ε, επιπτήσεων ε, για κάποιες χώρες της Μέσης Ανατολής. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε όλοι θεώρησαν ότι πρόκειται για πολλωστή φορά για μέτρα κατά της δημοκρατίας από τους φίλους μας, τον εντός εισαγωγικών φίλο μας τον κύριο Τραμπ, αλλά ε, την Τρίτη το Ενωμένο Βασίλειο ενέκρινε αντίστοιχους περιορισμούς. Πρόκειται για κάτι λοιπόν το οποίο συζητούν και οι υπηρεσίες σας αυτή τη στιγμή και ποια είναι η θέση του Επιτρόπου ε, για την κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Νάταλη. Η Γιούντιθ ε, από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα αν μου επιτρέπετε να κάνω μια σύγκριση, ένα παραλληλισμό μεταξύ της σημερινής εισαγωγή του Επιτρόπου για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και της πέμπτης έκθεσης προόδου για την ασφάλεια στην Ένωση. Στην έκθεση προόδου, που ήταν πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα, επισημάνατε την σπαστικοποίηση, πώς θα αντιμετωπίσουμε τους ε, ε, τζιχαντιστές που επιστρέφουν, ε, τους ε, εύκολους στόχους και είπατε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιες απειλές στην ασφάλεια έσωθεν απειλές και ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να προλάβουμε, να προβλέψουμε και να αποτρέψουμε αυτές τις εσωτερικές απειλές στην ασφάλεια. Ε, επίσης θέλουμε διασυνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων που όμως επικεντρώνονται κυρίως στις έξωθεν απειλές στην ασφάλεια. Και αυτό είναι προβληματικό. Για παράδειγμα, η Eurodac. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Πρόκειται ένα σύστημα που θέλει να επιτρέψει το Δουβλίνο να λειτουργήσει ε, και που κάνει τη διάκριση μεταξύ των ετούντων άσυλο και Τώρα θέλουμε να συμπεριλάβουμε στο σύστημα και επιστρέφοντες και να χρησιμοποιείται και σε δικαστικές έρευνες. Νομίζω ότι είναι ανησυχητική αυτή η επέκταση και τι γίνεται με την πιθανότητα παραποίησης των στατιστικών στοιχείων σε περίπτωση που αρχίζουμε και χρησιμοποιούμε τα ε, δακτυλικά αποτυπώματα και αρχίζουμε και βάζουμε στο σύστημα παιδιά εξάχρονα και το χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο για τις δικαστικές έρευνες. Μήπως ε, μετά από μια διετία θα έχουμε όλο και περισσότερα παιδιά ε, μετανάστες σε στατιστικές για, για στοιχεία εγκλημάτων μόνο και μόνο επειδή βρέθηκαν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα στο Eurodac, στο Eurodac και επειδή βρέθηκαν ε, ακριβώς σε αυτή τη χρονική περίοδο της διεύρυνσης ε, σε λάθος τόπο. Νομίζω ότι αντί να συσπηρώνουμε τις κοινωνίες μας, δημιουργούμε μία επιπλέον ανασφάλεια για τους μετανάστες που θέλουμε να τους εντάξουμε στην κοινωνία και όχι να τους περιθωριοποιήσουμε. Και η τελευταία ερώτηση που είχα υποβάλει και στην προπαρασκευαστική συνάντηση που είχαμε με τους εμπειρογνώμονες. Ερώτηση έκανα, αλλά απάντηση δεν έλαβα. Και θα ήθελα να αντιληφθούμε προς όλη αυτή η ενσωμάτωση, η ολοκλήρωση. Γιατί έχουμε ένα αστυνομικό που σταματά κάποιον και έχει μια τεράστια βάση δεδομένων. Μπορεί να βάλει μέσα ένα όνομα και να λάβει μια αίτηση παροχή πληροφοριών ή όχι. Κανένα όμω δεν μου απάντησε πώ λειτουργεί αυτό το σύστημα και τι σημαίνει όταν κάποιο κάνει το hit αυτό την αίτηση παροχή πληροφοριών ή δεν κάνει το hit. Στην προπαρασκευαστική συνάντηση με αστυνομικούς πριν από δύο εβδομάδες μου είπαν ότι είναι υπέρ της μεγαλύτερης διασυνδεσιμότητας, αλλά δεν βρέθηκε ούτε ένας να μου δώσει ένα παράδειγμα. Αυτό ζητούσε ένα απλό παράδειγμα για το πώς μπορεί κανείς έχοντας τα σωστά στοιχεία την κατάλληλη στιγμή να παρεμποδίσει ή να αποτρέψει μια απειλή. Θέλω παραδείγματα απτά για να καταλάβω αν είναι εφικτή τελικά αυτή η διαλειτουργικότητα. Ευχαριστώ κυρία Χολμάιερ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Αρχικά θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι αυτά τα κράτη, τα πέντε κράτη που δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει την απόφαση πριν. Γιατί πράγματι η μη εφαρμογή αυτής της ε, έκθεσης από τον Αύγουστο του 2011 ε, είναι μια πολύ μεγάλη περίοδος και ενδεχομένως να ε, ε, ε, λόγω μάλλον και της τρομοκρατικής απειλής που αντιμετωπίζουμε θα πρέπει επιτέλους να γίνει ε, η εφαρμογή αυτή. Τουλάχιστον επιτέλους ξεκίνησε η διαδικασία ε, επί παραβάση της συνθήκης γιατί εξ όσων γνωρίζω ε, δεν συνέβη κάτι τέτοιο ούτε το 2012 ούτε το 2013. Δεύτερον, μπορείτε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα όσον αφορά ε, τις εργασίες αυτής της ομάδας ε, εργασίας για την διαλειτουργικότητα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και το έργο της Επιτροπής αυτής και θα ήθελα η Κομισιόν να μας δώσει και κάποια παραδείγματα. Εγώ χθες άκουσα πολλά παραδείγματα στη συνδιάσκεψη της Ευρωπόλ όπου αναδείχθηκαν προβλήματα λόγω της έλλειψης της διαλειτουργικότητας των βάσεων δεδομένων των αστυνομικών αρχών, όπου πράγματι δημιουργούνται προβλήματα και δυσκολίες. Και εδώ, όπως είπε και η συνάδελφος τη ε, δημιουργούνται κενά ε, λόγω της ε, έλλειψης της απουσίας δεδομένων που πολλές φορές οφείλεται στην ε, μη επαρκή ανταλλαγή δεδομένων που υπάρχουν στη μία βάση δεδομένων. Πολλές φορές δηλαδή υπάρχουν πληροφορίες αλλά δεν ε, ανταλλάσσονται έγκαιρα με αποτέλεσμα να μην μπορούν ούτε να συγκριθούν ούτε να τεθούν σε υπεξεργασία έγκαιρα. Έπειτα έχω και ένα ερώτημα για την ανάλυση των δεδομένων. Χθε ε, στην, ε, στην, στην διάσκεψη αυτή που συμμετείχα άκουσα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί να γίνει ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων, των πληροφοριών. Αυτή η ανάλυση, ή μάλλον οι μονάδες, τα τμήματα ανάλυσης, μήπως θα έπρεπε να στελεχωθούν ακόμα περισσότερο προκειμένου να μπορούν να ε, παρέχουν σωστές και χρήσιμες πληροφορίες στην ε, ε, Ευρωπόλ, ώστε και η Ευρωπόλ, αλλά και όλες οι αστυνομικέ αρχές να μπορούν να επιτελούν σωστά το έργο τους. Ευχαριστώ, κυρία Τσινίτση. Κυρία Κινίτση, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε τον Επίτροπο για τη σημερινή του παρουσία. Εγώ ήθελα να είμαι παρούσα, για να καταλάβατε, ήμουν στη Ρώμη για την υπογραφή των 60 ετών, αλλά σήμερα ε, θεώρησα ότι ήταν και καθήκον, αλλά και ανάγκη να βρεθώ εδώ σήμερα. Και θα ήθελα καταρχάς να σας εκφράσω την αλληλεγγύη μου για τα θύματα της χθεσινής επίθεσης Πιστεύω ότι η προστασία των θυμάτων που συμπεριλάβαμε και στην οδηγία για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας ήταν και επικαιρή, αλλά χρειάζεται και περαιτέρω εφαρμογή και επιτρέψτε μου να το πω αυτό ε, σήμερα ειδικά ε, όσον αφορά το θέμα της συζήτησής μας. Ε, ε, αν όντω είναι αλήθεια και το απέδειξε και η χθεσινή επίπεδα ότι αυτές οι, επίθεση, ότι αυτές οι επιθέσεις συμβαίνουν εντελώς ε, τυχαία, ε, αλλά υπάρχουν ε, διασυνοριακά εγκλήματα, τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα και το είδαμε αυτό και στην οδηγία για την τρομοκρατία. Χρειάζεται αναγνω, συνεργασία και να αυξήσουμε το επίπεδο συνεργασίας. Ανταλλαγή πληροφοριών είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική στιγμή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μορφές εγκληματικότητας, για να μπορέσουμε να ε, προσφέρουμε και πάλι ασφάλεια στους πολίτες μας. Σας ευχαριστώ για την ευρύτερα και πληρόστατη παρουσίαση, παρά το γεγονός ότι ήσασταν συνοπτικοί, ε, συνοπτικός, συγγνώμη. Οι συνάδελφοι είπαν τα περισσότερα, αλλά θα ήθελα να πω και το εξή. Εσεί αναφερθήκατε σε ε, τμηματική πρόσβαση στο σύστημα VIS, στο γεγονό ότι κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα προσφορήσει σε αποφάσει προύμ ε, στην οδηγία για τα PNR, τα, τα στοιχεία ονομάτων επιβατών που ακόμα δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή και θα μπορούσα να πω κι άλλα, το SIS κλπ. Να ρωτήσω το εξή. διαπιστώθηκαν κάποιες ιδιαιτερότητες για κάποιες χώρες που ε, προσχωρούν και συνεισφέρουν στη διαβίβαση δεδομένων και κάποιες χώρες ε, δίνουν περισσότερα στοιχεία από ό,τι άλλες. Για κάποιες χώρες λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε πιο ουσιαστική προσχώρηση και κάποιες άλλες κάνουν πολύ περιορισμένη χρήση αυτών των εργαλείων. Για ποιον λόγο γίνεται αυτό κατά την άποψή σας και ε, ποιοι είναι οι μηχανισμοί και τα συστήματα για να μπορέσουμε να συμβιβάσουμε αυτές τις Επίση, Επίσης, οι συνάδελφοι επεσήμαναν τα θέματα της διαλειτουργικότητα και εγώ συμφωνώ λίγο με τις ε, ανησυχίες που εκφράστηκαν και το γεγονό ότι θα πρέπει ε, να δράσουμε γέρος από αυτών των ε, στοιχείων. Και το είπε προηγουμένως και η κυρία Χολμάιερ, πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο interface για πρόσβαση στα δεδομένα, γιατί ξέρουμε ότι τα συστήματα αυτά είναι σίγουρα αποτελεσματικά και απαραίτητα, αλλά ορισμένες φορές ε, για τους χρήστες ε, που, που καταχωρούν τα στοιχεία, που θέλουν να λάβουν κάποιες πληροφορίες μέσω αυτών των βάσεων δεδομένων, το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο interface ε, δημιουργεί αρκετά προβλήματα και να αναφερθώ ακροθυγός και σε κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι της παρούσης αυτή τη στιγμή, αλλά το αναφέρατε εσείς και το είπε και η κυρία Γκρισμέκ προηγουμένως, το θέμα της αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος. Το ξέρω ότι δεν είναι αποκλειστική ε, η σχέση του με το θέμα που συζητούμε σήμερα, αλλά πιστεύω ότι το κυβερνοέγκλημα είναι ε, μια μορφή εγκλήματος που δεν είναι επικίνδυνη μόνο για κάποιον πολίτη ε, που συνδέεται στο διαδίκτυο, αλλά μπορεί να έχει και πάρα πολύ σημαντικού κινδύνους και για κυβερνήσεις και για κράτη. Μήπως θα μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε κάτι παραπάνω και για το θέμα αυτό. Ε, ούτως ή άλλως και αυτό είναι θέμα ασφαλείας και πρέπει να παρέμβουμε διότι αφορά και την ασφάλεια των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Κινίτση. Ο κύριος Κουέλιο τώρα. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον Επίτροπο που ήρθε. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω, όπως και οι συνάδελφοι, την αλληλεγγύη μου προς εσάς και τους συμπατριώτες σας αυτή τη στιγμή του πένθους. Και όπως είπατε, εδώ εξετάζουμε τα υφιστάμενα συστήματα, δηλαδή τις ήδη ισχύουσες βάσεις δεδομένων. Γι' αυτό και πιστεύω ότι αυτό πρώτα θα πρέπει να κάνουμε, να εξετάσουμε τα υφιστάμενα εργαλεία που έχουμε συμφωνήσει να τα εφαρμόσουμε επιτέλους και μετά να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Και περιμένω την έκβαση της ομάδας υψηλού επίπεδου για τη διαλειτουργικότητα που θα αποτελέσει σημείο αφετηρίας και για περαιτέρω συζητήσεις. Πάντως θα ήθελα να επισημάνω ότι οι περαιτέρω δράσεις για τη διαλειτουργικότητα ή την στρατηγική διαχείριση ή επεξεργασία πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μετά την έγκριση ή απόρριψη των συστημάτων που ήδη έχουμε ενισχύει. Και όπως είπατε κι εσείς ε, από την αρχή την ανάλυση των καθηκόντων σας, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας είναι να βελτιώσουμε και να εφαρμόσουμε αυτά που ήδη έχουμε. Αναφέρθηκε το σύστημα πληροφοριών Schengen. ΣΥΣ, ε, καλό παράδειγμα εφισταμένου ε, εργαλείου που ε, σταδιακά, ε, τακτικά μάλλον αξιολογείται και βελτιώνεται. Μάλιστα είμαι ο εισηγητής για το θέμα αυτό και πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε και στη συνέχεια. Και μάλιστα με ταχύς ρυθμούς. Συμφωνώ με το σχόλιο σας για τα δακτυλικά αποτυπώματα. Τα βαριμετρικά στοιχεία ήδη υπήρχαν από το ΣΥΣ 2 και δεν αξιοποιήσαμε αυτή τη νομική διάταξη του δεύτερου συστήματο πληροφοριών Σέγγεν. Και τώρα, όχι μόνο για την αποθήκευση δεδομένων, αλλά και για τι διαδικασίε υποβολής ετοιμάτων, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων. Αναφέρθηκε τώρα η αποφάση PRIM και το σύστημα PNR. Ε, ε, ζητήσατε συνοπτική διαδικασία και άμεση ε, εφαρμογή του PNR και ένα χρόνο μετά ούτε οι μισές μέλη δεν το έχουν εφαρμόσει. Σε ό,τι αφορά ε, την απόφαση πριν. Εννέα χρόνια μετά την έγκριση αυτής της απόφασης και έξι χρόνια μετά την εκπνοή της περίοδου εφαρμογής, πέντε κράτη-μέλη εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν και να μην συμμορφώνονται με την απόφαση αυτή. Και μάλιστα το Συμβούλιο δεν δίνει καν στατιστικά στοιχεία για τη χρήση της απόφασης πριν. Και τέλος, είμαι ήμουν ανέκαθεν υπέρ τη καλύτερη ανταλλαγής πληροφοριών και όχι αύξηση των πληροφοριών. Η Ευρωπόλ έχει ε, πολλές αρμοδιότητες σχετικά. Και μάλιστα αυξάνονται, ε, η, αυξάνεται αποστολή στοιχείων προς την Ευρωπόλ. Ερωτώ λοιπόν, τα κράτη-μέλη όντως προσφέρουν καλύτερες πληροφορίες στην Ευρωπόλη, απλώς ε, αδιάκριτα στέλνουν όλες τις πληροφορίες, οπότε αυξάνεται έτσι ο όγκος τεχνητά, χωρίς όμως ποιοτική διάκριση. Ευχαριστώ. Η Σόφη Ιντβελτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που έχουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα, γι' αυτό και παρίσταμε εδώ. Είναι ε, πιο επίγουσα από ποτέ αυτή η συζήτηση. Είμαστε όλοι πολύ θλιμμένοι αλλά και πολύ θυμωμένοι με τα χθεσινά γεγονότα διότι ακούμε ότι το Ισλαμικό κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές όπως κάνουν πάντοτε βεβαίω στους τελευταίους μήνες. Υπάρχουν διάφοροι ε, μεμονωμένοι ε, άτομα τα οποία πιστεύουν ότι είναι ήρωες ενώ στην πραγματικότητα πλανώνται, πλάνιν. Και χθε μάλιστα είχαν τα πιο απλά αντικείμενα που μπορεί κανείς να έχει ένα αυτοκίνητο και ένα μαχαίρι. Είναι πραγματικά αξιολύπητοι οι άνθρωποι αυτοί, αλλά παρόλα αυτά είναι σε θέση και προκαλούν πολύ μεγάλη ζημιά. Και κάθε φορά ακούμε το ίδιο ρητό, ότι δεν θα επιτρέψουμε σε αυτό το γεγονός να αλλάξει τον τρόπο ζωή μας και ταυτόχρονα αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους να ε, ε, θέτουν υπό αμφισβήτηση και το κράτος δικαίου μας και τον τρόπο ζωή μας. Και αυτό γίνεται εδώ και 15 χρόνια. Είπατε για το κλείσιμο των κενών. Φυσικά κανείς δεν πρόκειται να διαφωνήσει με αυτό, αλλά τι ακριβώς σημαίνει ένα τέτοιο σύνθημα. Εγώ φυσικά με τα χαράς ε, θα υποστηρίξω ε, οποιοδήποτε σύστημα βελτίωσης της ανταλλαγής των πληροφορών Είμαι και ε, υπέρ της υποχρεωτικής μάλιστα ανταλλαγής πληροφοριών. Αλλά τι συγκεκριμένα θα κάνουμε. Αν δούμε τη χθεσινή επίθεση, ο άνθρωπος αυτός γεννήθηκε στην Βρετανία, ήταν γνωστός στην, στις μυστικές υπηρεσίες και ήταν γνωστό ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί, ήταν εξτρεμιστής σε πάση περιπτώσει, όπως θέλετε πείτε τον. Και και σε τι μας βοήθησε τελικά αυτός. Σε κάθε επίθεση που έχει γίνει στην επικράτεια της ε, Ένωσης από την 11η ε, Σεπτεμβρίου και έπειτα, γνωρίζουμε τέτοιου είδους πληροφορίες εκ των προτέρων. Και κάθε φορά τι κάνουμε, ζητούμε ακόμα μεγαλύτερη συλλογή πληροφοριών, ακόμα περισσότερων πληροφοριών. Το πρόβλημα είναι πώς οι πληροφορίε αυτές που ήταν διαθέσιμες για αυτό το άτομο, πώς θα καταφέρουμε τέτοιου είδους πληροφορίε να τις ε, αξιοποιήσουμε ή πώς μπορούν να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί κάποια στιγμή να ξυπνήσει, να πάρει ένα μαχαίρι και να σκοτώσει κόσμο. Χθες ε, ε, έγινε ε, κάτι αντίστοιχο και στην, στην, στην ε, ε, Αμβέρσα. Δηλαδή είδα έναν άνθρωπο να, να, να τρέχει με πολύ ψηλή ταχύτητα μέσα στους δρόμους. Μπορεί να ήταν τρομοκράτης, μπορεί και όχι. Γεγονός είναι ότι πώς, πώς, είναι, πώς είναι δυνατόν να ό,τι πληροφορίες και αν συλλέξουμε δεν πρόκειται να τους βρούμε αυτούς όσες πληροφορίες και να συλλέξουμε. Χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Όταν αναλάβατε τα καθήκοντά σας μιλήσατε πολλά για, τις, για την άλλη πλευρά, για την πρόληψη, για τις κοινωνικές διαστάσεις κτλ. κτλ. Τι κάνει λοιπόν η Κομισιόν σε αυτό το μέτωπο. Για το PNR. Δεν, δεν θέλω να σας πω ότι σας τα έλεγα, αλλά σας τα έλεγα. Πέρσι είχαμε την ψηφοφορία, εγώ είχα καταψηφίσει, γιατί ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι ακριβώς η, ίδια λογική με τα όσα είχαμε στην περίπτωση της ε, αποθήκευσης δεδομένων, της δεδομένων δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια. Είναι ηλίθιο αυτό το πράγμα. Τι κάνει η Κομισιόν λοιπόν, το συζητήσαμε την, τελευταία φορά, μας είχατε υποσχεθεί ότι θα μας δώσετε μια γραπτή ενημέρωση σχετικά και, και συμπεριλαμβανομένων και των δημοσιονομικών πτυχών, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει 130 ε, εκατομμύρια ευρώ για αυτό το PNR. Ε, θέλω να ξέρω τι, που, που πήγαν αυτά τα λεφτά. Τελευταίο ερώτημα. Μιλήσατε για τη Γαλλία και την συγχαρήκατε που δεν ακύρωσε τη διοργάνωση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Συμφωνώ απολύτως, αλλά ε, ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν την ε, ε, κατάσταση έκτακτης ανάγκης η οποία εξακολουθεί να ισχύει στη Γαλλία. Είναι αιτιολογημένο κάτι τέτοιο ή θα αρχίσουν και άλλες χώρες να ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Γιατί ε, ε, ακούμε πολλά για τη διατήρηση του δικού μας ε, τρόπου ζωής κτλ. Ε, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν μπορεί παρά να είναι εκ, αυτό που λέει και, η λέξη έκτακτης ανάγκης και όχι μια μόνιμη κατάσταση. Ευχαριστώ. Η Μάριου Λαουρεστίν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συνεχίσω αυτά που είπε αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες. Είναι κάπως περίεργη η κατάσταση. Όταν μιλούμε για προστασία δεδομένων, όλοι ε, ανησυχούμε γιατί οποιοδήποτε θα μπορούσε να είχε εντοπιστεί, να, να καταρτιστεί το προφίλ του παντού και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή τη βαθύτατη ανησυχία. Και εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που ήταν συσημασμένο ε, και ήταν γνωστό για πολύ καιρό και παρόλα αυτά το προφίλ του δεν ήταν έτοιμο, δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν και ήταν ε, απροσδόκητο να εμφανιστεί εκεί που εμφανίστηκε και να διαπράξει αυτό που έκανε. Και έχουμε μια τεράστι... ένα τεράστιο κενό μεταξύ των δύο αυτών καταστάσεων. Επίση, ε, έχουμε και το θέμα τη ποιότητα τη ανάλυση των δεδομένων. Όχι μόνο των βάσεων μαζικών δεδομένων, Θέλουμε ποιοτική επεξεργασία δεδομένων ό,τι αφορά την κατάρτιση προφίλ. Με τη θετική έννοια, όταν χρησιμοποιούμε το profiling για να αποτρέψουμε τέτοιου είδους επιθέσει. Επίση, επιθέσεις. Επίσης, τι γίνεται με τους πόρου που αφιερώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να βοηθήσει ε, τους ερευνητές, ώστε να έχουμε την τελευταία λέξη της έρευνας και της τεχνολογίας και της δημιουργίας γνώσης και των νέων μεθοδολογιών γιατί πρόκειται για μία μελέτη, μία, ένα τομέα υψηλής ειδίκευσης. Εμείς είμαστε πολιτικοί και μπορούμε να μιλάμε για χιλιάδες ώρες και να μην συμβαίνει τίποτα, γιατί δεν θα έχουμε κατάλληλους εμπειρογνώμονες, ώστε να κάνουν αυτές τις ποιοτικέ αναλύσεις και να δημιουργήσουν και συστήματα, γιατί τα συστήματα δεδομένων συστήματα είναι. Δεν είναι απλώς ένα τεράστιο καλάθι δεδομένων. Και αυτή τη γνώση θέλουμε γίνεται βελτίωση των συστημάτων. Ποιοτική βελτίωση, όχι ποσοτική. Υπάρχει βελτίωση στον τρόπο ανάλυσης των δεδομένων. Γιατί ε, οι αρχές επιβολής του νόμου, οι αρχές ασφαλείας εκπαιδεύονται δεόντως, καταρτίζονται επαρκώς. Γιατί είπαμε ότι πολλές χώρες ε, γιατί πολλοί, ακόμη και είναι στο σύστημα, δεν ξέρουν πώς να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα. Δεν εμπιστεύονται τα δεδομένα, δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεν έχουν και την πνευματική ικανότητα να τα αξιοποιήσουν. Πώς θα επιτύχουμε λοιπόν σε διανοητικό επίπεδο βελτίωση για να γίνεται αξιοποίηση αυτό το δεδομένο ώστε να ενισχύεται πραγματικά η ασφάλεια. Και στην πατρίδα μου έχουμε αυτό το κέντρο ασφάλειας των δεδομένων, αναφέρεται και το Λίσσα, ποιος θα είναι ο ρόλος αυτού του κέντρου. Ε, μπορεί να γίνει ένα κεντρικό, τέτοιο συντονιστικό κέντρο η Λίσσα για την ασφάλεια των δεδομένων. Κυρία Χολμάιερ. Ένα θέμα ήθελα να αναφέρω μετά την ε, Σόφη Ίντβελ. Νομίζω ότι ως Επιτροπή ΛΥΜΠΕ δεν πρέπει να υιοθετήσουμε τον ρόλο του κατηγόρου Αντιθέτως, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε πολλά κράτη-μέλη έχουν, επίσης αποτραπεί επιθάσεις, έχουν ανταλλαχθεί πληροφορίες, έχουν διαβιβαστεί σωστές και έγκαιρες πληροφορίες και αυτό που έγινε στην Αμβέρσα όπου ε, ε, ε, ε, ευρέθησαν από τις αστυνομικές αρχές και όπλα και πυρομαχικά. Ε, φαίνεται δηλαδή να πρόκειται για μια περίπτωση αποτροπής τρομοκρατικού χτυπήματος και σε αυτή την περίπτωση πράγματι πρέπει να αναγνωρίσουμε στην αστυνομία της Αμβέρσας ότι πράγματι έδρασε έγκαιρα και γρήγορα. Όσον αφορά ε, το περιστατικό στο Λονδίνο, δεν μπορούμε να αποδίδουμε την, ε, την ευθύνη ε, για τέτοιου είδου περιστατικά στο γεγονό ότι συλλέγονται πληροφορίε. Το PNR, για παράδειγμα, δεν είναι ένα εργαλείο μόνο για την καταπολέμηση τροποκρατία, ούτε το είπε ποτέ κανεί αυτό. Είναι μία μέθοδο, είναι ένα δομοστοιχείο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο, είναι ένα εργαλείο για την καταπολέμηση και τη τρομοκρατία και περιμένω από τα κράτη-μέλη να το προχωρήσουν όπως το έχουν κάνει και στο παρελθόν με άλλα θέματα. Και νομίζω, ε, κύριε Επίτροπε, είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο να αναδειχθούν ορισμένες φορές και ορισμένα επιτεύγματα. Πράγματα που έχουν επιτευχθεί θετικά. Γιατί ε, ε, θα ήταν πολύ χρήσιμο να μάθουμε για παράδειγμα ποια χτυπήματα ή ποιες επιθέσεις απετράπησαν χάρη στο PNR. Γιατί συνήθως ακούμε στις ειδήσει για τις, ε, για τις ελλείψεις, για τα προβλήματα, για τις δυσκολίες, για την έλλειψη διαβίβασης πληροφοριών κτλ. κτλ. Αλλά εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποια θετικά επιτυγχάνονται χάρη στα μέσα και στα εργαλεία που έχουμε ε, συστήσει. Κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι η κυρία Χολμαϊέρ αποδέχεται ότι έχουμε ελευθερία του λόγου σε αυτή την Ήπειρο και μπορώ κάλλιστα να πω την άποψή μου. Βεβαίω, βεβαίω, λέει ο Πρόεδρο. Ε, να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα και να πω ότι κάποια από αυτά τα θέματα, η πρόληψη για παράδειγμα, ένα από τα σοβαρά πράγματα που αναφέρθηκαν εδώ είναι για το κατά πόσο μπορούν να προλάβουμε αυτές τις επιθέσεις. Η Επιτροπή μας ασχολείται, έχει κάνει πολλή δουλειά, ξέρετε, είχαμε και όλα αυτά τα θέματα με τις μαζικές παρακολουθήσεις, έχουμε προλάβει αρκετές επιθέσεις, αλλά Αυτά είναι θέματα τα οποία ανακύπτουν σε διάλογο για την ασφάλεια. Ε, κάποια πράγματα τα έχουμε προλάβει, αλλά δεν γνωρίζουμε και πολλά, γιατί τα περισσότερα είναι μυστικέ πληροφορίε τι οποίε δεν δημοσιεύουμε ε, στο ευρύ κοινό. Ε, θέματα λοιπόν για το διάλογο ασφαλείας είναι θέματα τα οποία βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα και υπάρχει ε, και νομική δυνατότητα. Το PNR, η ε, προθεσμία είναι το 2019 και κάποια κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα ακόμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένα σύνθετος τομέας αυτό στον οποίο υπάρχει πρόληψη. Υπάρχουν και άλλα θέματα όμως. Και πρέπει να τα φύγουμε αυτά τα ζητήματα κατά την άποψή μου. Δεν ε, έχω κανένα πρόβλημα να τον ακούγονται όλες οι απόψεις. Τι τα λέω τώρα λεφτά; αυτά. Προσπαθώ να κάνω το διαμεσολαβητή όταν δεν υπάρχει καν λόγο. Τι τα είπα. Ε, ε, ε ένα λεπτό χαμένο δεν θα αλλάξει τίποτα. Προσπαθώ να διαμεσολαβήσω ανάμεσα στη Σόφη Ινέτβελτ και την κυρία Χολμάιερ. Δεν ξέρω αν υπήρχε λόγο που ανακατεύτηκα. Τέλος πάντων, πέμπτη απόγευμα ήταν δύσκολη εβδομάδα. α το πάρουμε απόφαση. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση όμως ε, να μειώσω την αξία του σχολείου αυτού για την πρόληψη των επιθώσεων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σχόλιο. Λοιπόν, γιατί σα ευχαριστώ που είστε εδώ. Γιατί είναι πέμπτη απόγευμα. Αλλάξαμε το πρόγραμμα. Κάποιοι πήγαν στην προπαρασκευαστική συνεδρίαση. Ε, υπήρχε πρόβλημα ε, στον προγραμματισμό. Άλλαξε το πρόγραμμα της ε, η Επιτροπή. Καταφέραμε λοιπόν να κάνουμε αυτό το διάλογο γιατί ο κόσμο άλλαξε το πρόγραμμά του για να είναι εδώ σήμερα. Σα ευχαριστώ λοιπόν που είσαστε εδώ σήμερα. Κύριε Επίτροπε, έχετε ένα μακρύ κατάλογο θεμάτων, αρκετά θέματα που αφορούν εφαρμογή και το ETIAS όμως και άλλα θέματα και έγιναν και αρκετές συζητήσεις αυτή την εβδομάδα. Συζητήσαμε το ETIAS ε, μεταξύ άλλων. Σας παρακαλώ λοιπόν κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να μας απαντήσετε σε όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ενδιαφέρεστε τόσο για αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ και για την ελεγγύη μετά από τα πιο πρόσφατα ε, θλιβερά ε, γεγονότα σε αυτή τη θλιβερή σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο το δυνατόν περισσότερε ερωτήσει. Αν νιώσετε κάποια στιγμή ότι δεν σα απάντησα, να μου το πείτε. Αν δεν απάντησα γιατί δεν ξέρω την απάντηση, θα σα το πω και θα σα ε, στείλω απάντηση γραπτό. Πρώτον, πώς θα ε, δομήσω την απάντησή μου. Όπως είπε ο κύριος Κοέγιο, μεταξύ άλλων, το βασικό θέμα που εξετάζουμε σήμερα είναι τι γίνεται με τα συστήματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Και πολλοί από εσά ε, ε, επικεντρώθηκαν σε αυτά, όπως και εγώ στα σχόλιά μου, και επομένως θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτά που θίξατε. Κάποιοι από εσά και δικαίω κατά την άποψή μου, ε, πήγατε το θέμα λίγο ευρύτερα γιατί κάνουμε ένα διάλογο ασφαλεία. και ε, θέσατε θέματα ε, για τη διαλειτουργικότητα και τη σχέση μεταξύ διαλειτουργικότητας και των συστημάτων που έχουμε στη διάθεσή μας και θέματα που αφορούν την ευρύτερη διαλειτουργικότητα. Θα απαντήσω και σε αυτά, αλλά σημειώνω ότι πρέπει να επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό. Κάποιοι από εσά έθιξαν θέματα πρόληψης. Υπό την έννοια της αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης και ε, της προώθησης καλών σχέσεων μεταξύ ε, μιας κοινότητας και να μπορέσουμε να βρούμε και σημεία συνάφειας μεταξύ των κοινοτήτων μας. Η κυρία Σαρχεντίνη αναφέρθηκε σε αυτό. Ε, δεν θα ήθελα ε, να τα αποφύγω αυτά τα θέματα σε καμία περίπτωση. Ε, τα συζητήσαμε, όπως επεσήμανε κάποιο σε μία από τις πρόσφατες εκθέσεις πρόοδου για την ασφάλεια στην Ένωση. Εγώ τα συζητώ τα θέματα αυτά και μάλιστα τα συζήτησα και χθε σε μία ε, ε, παρουσίαση βιβλίου για τη ριζοσπαστικοποίηση. Ε, αν θέλετε μπορείτε να βρείτε και τις παρατηρήσεις μου στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με τη ριζοσπαστικοποίηση και τι μπορούμε να κάνουμε στις κοινότητές μας και αν θέλετε να κάνουμε ξεχωριστή συνεδρίαση εις βάθος για τα θέματα αυτά, ευχαρίστως ε, να προσέλθω. Κάποιοι από εσά, η κυρία Ίνετφελτ ε, τελευταία, ρώτησαν με διαφορετικό τρόπο τι διδάγματα αντλούμε από τις διάφορες επιθέσεις που συμβαίνουν. Προσπαθούμε να μάθουμε από τις επιθέσεις και δεσμευόμαστε από αυτού, το συζήτησα και έγραψα και από αυτού και, την περασμένη εβδομάδα μάλιστα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μπορέσουμε σίγουρα να αποτρέψουμε μελλοντικές επιθέσεις. Κάποιες εξ αυτών των επιθέσεων, ειλικρινά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις προλάβουμε. Ιδιαίτερα αν πρόκειται για κάποιον ο οποίος ακόμα και σε κάποια στιγμή μπορεί να ε, προσέξε, προσέλξε το ενδιαφέρον των αστυνομικών αρχών ή άλλων. Όλοι όσοι βρίσκονται στο στόχαστρο αυτών των υπηρεσιών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ανα πάσα στιγμή ε, είναι στο στόχαστρο. Ε, ο καθένας ενδιαφέρεται, ε, αξιολογούνται κάποιοι άνθρωποι ε, για το κατά να αποτελούν κίνδυνο ή όχι. Και υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις τις οποίες κάποιος ε, ε, ήταν άτομο ενδιαφέροντος και μπορεί να έχει βρεθεί πιο κάτω στον κατάλογο και μετά επειδή προέκυψε κάποιον επεισόδιο ταχύτητα της ριζοσπαστικοποίησης μπορεί να κάνει μια επίθεση. Και το έχουμε δει κάτι τέτοιο και κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε κάτι αντίστοιχο και στο μέλλον. Κάποιος λοιπόν ο οποίος μόλις ριζοσπαστικοποιήθηκε ή ξανά ριζοσπαστικοποιήθηκε ε, και επιτίθεται με ό,τι έχει στη διάθεσή του για να ε, μπορέσει να διαπράξει την επίθεση και το οργανώνει και μόνος του ε, δεν έρχεται σε επαφή σε κάποιο, με κάποιο ευρύτερο δίκτυο, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει ανησυχία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και όταν Αναφερόμαστε στα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από κοινού, προκειμένου να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την ασφάλειά μας. Νομίζω ότι είναι απόλυτα σημαντικό να μην δώσουμε και λανθασμένη εντύπωση ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να εξαφανίσουμε όλου του κίνδυνου. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και δεν υπάρχει μηδενικό κίνδυνος. Ε, αυτό σημαίνει ότι είναι λάθος να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ρεαλιστική αξιολόγηση και να δράσουμε εκεί που μπορούμε. Όχι, ε, νομίζω ότι ε, αυτό περιμένει ο κόσμος από εμά και νομίζω ότι αυτό είναι και αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε όλοι από κοινού. Εγώ ε, είμαι υπέρμαχος μιας αποτελεσματικής αξιολόγησης, θα γίνει αξιολόγηση, θα ε, την έχουμε και αργότερα μέσα στο καλοκαίρι αυτή την αξιολόγηση και ελπίζω τότε να είναι ε, μία εκ των διαφόρων ανταλλαγών που θα έχουμε μετά από τη δημοσίευση της αξιολόγησης. Ε, προφανώς και δεν θα είναι τέλεια για όλους σας, αλλά θα είναι μια απόπειρα έστω να εμβαθύνουμε τη συζήτηση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουμε λάβει τμήμα αυτού, προφανώς και αρκετοί από εσάς το αναφέρατε, είναι η βασική πρόκληση της εφαρμογής των μέτρων. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη ε, τα θέματα εφαρμογής. Το PNR, ε, το μητρό όνομα των επιβατών, είναι ένα εκ των παραδειγμάτων που ανέφεραν αρκετοί από εσά Υπάρχει ένα σχέδιο εφαρμογής, ε, σας το ε, κοινοποιήσαμε. Νόμιζα ότι σας είχαμε δώσει και κάποιες πληροφορίες για τη χρηματοδότηση. Εάν δεν έγινε αυτό ή σας οφείλουμε μια ενημέρωση, θα τα κοινοποιήσουμε και αυτά γιατί δεν κρύβουμε τίποτα. Γίνονται τα πάντα με πλήρη διαφάνεια, ε, και το τι κάνουμε με τα επιπλέον 20 εκατομμύρια που βρήκαμε φέτο για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη που χρειάζονται επιπλέον βοήθεια. Εάν υπάρχουν άλλα στοιχεία εφαρμογής τα οποία θα θέλετε ε, να εξετάσουμε περαιτέρω, είμαστε στη διάθεσή σας. Ε, Τζούλιαν, για το PNR νομίζω η προθεσμία είναι το 2019. Ναι, είναι την άνοιξη του 2018. Α, νωρίτερα ακόμα. Η ανησυχία που κατάλαβα εγώ είναι ότι ε, προχωράμε τόσο αργά προς αυτή την προθεσμία που οι συνάδελφοι ανησυχούν και αυτό έλεγε και η έκθεση. Δεν διαφωνώ σε καμία περίπτωση. Επίσης, ε, περιμένουμε τη Δευτέρα τους Υπουργούς ε, της Γερμανίας και της Γαλλίας, ε, Υπουργούς Εσωτερικών και θα θέσουμε και σε αυτό το θέμα. Μα δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας. Μακάρι να προχωρούσαμε ταχύτερα, και αν μπορείτε να με βοηθήσετε να συνεχίσουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για το θέμα αυτό, θα σήμαν ιδιαίτερα σε ευγνώμων. Εκεί που διαφωνώ κάπως με μερικούς από εσάς είναι ότι ακριβώς επειδή κάτι είναι δύσκολο στην εφαρμογή, δεν σημαίνει ότι ήταν λάθος η θέσπισή του. Γιατί μερικά από τα συστήματα αυτά πραγματικά είναι πολύ δυσεφάρμοστα σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ήταν άχρηστα ή ότι ήταν λάθος ο στόχος μας. Η απόφαση πριν συνιστά μια ιδιάζουσα πρόκληση και την αντιμετωπίζουμε με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Δεν προσπαθούμε να αποκρύψουμε τίποτα για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει και έχουμε δώσει και γραπτές πληροφορίες για το στάδιο της, των διαδικασιών υπεραβάση που γίνονται εις βάρος Ελλάδας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας και Κροατίας. Αυτές είναι οι πέντε χώρες για τις οποίες έχουν κινηθεί οι διαδικασίες. Και οι πέντε χώρες μας έχουν στείλει τις απαντήσεις, τις επεξεργαζόμαστε. Ε, δείχνουν οι απαντήσεις αυτές διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας ό,τι αφορά την, ε, την εφαρμογή της απόφασης πριν και αν υπάρχει ανεπαρκής ετοιμότητα ή τεκμήρια για την σοβαρή προσπάθεια εφαρμογής, θα περάσουμε στο δεύτερο, επόμενο στάδιο των διαδικασιών επί παραβάση. Αυτά λοιπόν ήταν τα θέματα που ξεπερνούσαν το αντικείμενο της σημερινής ε, συζήτησης που ήταν τα υπάρχοντα όργανα. Αλλά έκρινα σκόπιμο να το αναφέρω και αυτό. Και το ΕΦΙΣ ήταν τμήμα της, ε, το πιλωτικό πρόγραμμα ΕΦΙΣ. ΕΦΙΣ. θα είναι ανοιχτό σε όλα τα κράτη-μέλη, ελπίζω το συντομότερο δυνατό, γιατί υπάρχει η νομική βάση για αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, για την αυτόματη αναγνώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων και ε, βρήκα τα έξι κράτη που συμμετέχουν στο πιλωτικό αυτό πρόγραμμα. Είναι η Αυστρία, η Γερμανία, οι κάτω χώρες, η Πορτογαλία, η Λετωνία και η Ελβετία ως συνδεδεμένο κράτος. Για το πρόγραμμα ΕΤΙΑ, το σύστημα πληροφόρησης και αδειών ταξιδίου. Κατάλαβα ότι σε ενοχλεί κάπως ε, αυτή, αυτό το θέμα της ε, αξιολόγησης επιπτώσεων, αλλά δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι πάντα θα έχουμε εκτενείς ε, μελέτες επιπτώσεων, ανάλογα με τις προτεραιότητες και το τι επήγει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, την περίπτωση του αιτίας, ε, στηρίξαμε την πρότασή μας σε μια μελέτη σκοπιμότητας που είναι 280 σελίδων και μάλιστα τη δημοσιεύσαμε παράλληλα με την πρόταση. Ε, στη μελέτη ε, σκοπιμότητας έγινε ανάλυση των πιθανότητων και του αντικτύπου, αλλά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως πλήρης έκθεση ε, η μελέτη επιπτώσεων ή αντικτύπου. Ήταν περισσότερο σκοπιμότητας. Πάντως, πολύ ευχαρίστως να συνεχίσουμε τις επαφές ή κατηδίαν στην Επιτροπή, να συνεχίσουμε τις συζητήσεις κάποια άλλη στιγμή για τα τεκμήρια που συγκεντρώσαμε, τα σενάρια που διερευνήσαμε. Αν σας εξυπηρετεί, φυσικά σας, σας ενδιαφέρει. Από ό,τι ξέρω, στις αρχές Απριλίου θα γίνει μια συζήτηση μεταξύ των σκιωδών εισηγητών. Ίσως εκεί θα ήταν ευκαιρία να αναπτύξουμε το θέμα περισσότερο. Και όπως είπα και στην αρχή, Φαίνεται ότι όλοι τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι το θέμα είναι κατεπήγον, γιατί το ΕΤΙΑΣ είναι ένα από τα ζητήματα προτεραιότητας, όπως φαίνεται και στην κοινή διοργανική διακήρυξη. Σε ό,τι αφορά την ομάδα υψηλού επίπεδου, και το πώς θα συνδυαστεί αυτό το έργο της ειδικής αυτής ομάδας με τα υπάρχοντα συστήματα, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το επόμενο βήμα θα είναι η δημοσίευση της τελικής έκθεσης, οριστικής έκθεσης ομάδας υψηλού επίπεδου που θα υποβληθεί στις αρχές Μαΐου και κατόπιν θα υποβάλουμε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πιο συγκεκριμένες προτάσεις που θα αποτελέσουν τη βάση για τη συζήτηση μέχρι τα μέσα Μαΐου. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν μείζονες εκπλήξεις, γιατί συνεχίζονται οι συζητήσεις για το θέμα αυτό και μάλιστα πολύ με ρωτήσατε σήμερα το απόγευμα για κάποιες πτυχές της ε, ομάδας υψηλού επίπεδου, όπως το ενιαίο σημείο διαπαφής, το κοινό αρχείο ε, και αυτό δείχνει ότι έχουμε κάποια ιδέα για την πιθανή έκβαση της ομάδας υψηλού επίπεδου. Πάντως θα υποβληθεί, η ε, οριστική έκθεση και θα ακολουθήσουν προτάσεις. Πρόκειται για την αφετηρία μιας κοινή συζήτηση των τριών θεσμικών οργάνων για τη μελλοντική μας πορεία. Και μία από τις πιθανές ιδέες θα απαιτούσε ίσως και νομοθετικές αλλαγές. Αντί αυτή περίπτωση θα ακολουθεί η διαδικασία και στόχος για τη συζήτηση είναι να καταλήξουμε σε κοινή συνεννόηση για την ε, ακολουθητέα στρατηγική, προκειμένου η διαχείριση των δεδομένων για την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο αποδοτική και αποτελεσματική, με πλήρη σεβασμό των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και κατόπιν θέλουμε να συνεργαστούμε στην εφαρμογή αυτού του δικού χάρτη της κοινή στρατηγικής, με το χρόνο που χρειάζεται φυσικά για τη συζήτηση. Επίσης, σίγουρα θα εξετάσουμε από κοινού τον οδικό χάρτη και θα συνεργαστούμε για τη διαμόρφωσή του. Και επίσης θα ήθελα να τονίσω κάτι που τόνισαν ιδιαίτερα ο κύριος Κέλλερ και άλλοι, ότι θα πρέπει πρώτα να διεκπαιρεώσουμε τις εκκρεμείς υποθέσεις και εκ παραλίλου να οργανώσουμε συζήτηση για το μελλοντικό σχέδιο δράσης για την διαλειτουργικότητα. Δεν είναι ότι θέλω τέτοια συζήτηση, αλλά η εφαρμογή του σχεδίου εργασίας για την διαλειτουργικότητα θα πρέπει να ακολουθήσει την διεκπαιρέωση πρώτα των εκκρεμουσών υποθέσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι και το λογικό. Τώρα, τι σημαίνει αυτό. Αν συμφωνήσουμε το πρόγραμμα για τη διαλειτουργικότητα και ανακαλύψουμε ότι χρειάζονται κάποια νομοθετικά μέτρα για αναθεώρηση επιμέρους ε, θεμάτων, είτε που έχουν διεκπαιρεωθεί είτε που συζητούνται, και αυτό δεν είναι απίθανο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το σύστημα πληροφοριών Schengen. δεν έχουμε εδώ κάποια ρηξικέλευθη μεθοδολογία η διαδικασία. Νομίζω ότι αυτός είναι ο πιο επικοδομητικός τρόπος για την περαιτέρω μας πορεία. Ε, και θίξατε και κάποια άλλα ζητήματα. Επειδή δεν θέλω να μακρηγορήσω, ίσως δεν τα σχολιάσω όλα σήμερα λεπτομεριακά. Μερικά αφορούν και το θέμα της διαλειτουργικότητας, οπότε σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Το θέμα της ποιότητας των δεδομένων και η εισαγωγή των δεδομένων, αλλά και η ε, ποιότητα της ε, επεξεργασίας των δεδομένων και της ανάλυσης των δεδομένων είναι πολύ σημαντικά θέματα και θα εξετάσουμε στο μέλλον κάποιες προτάσεις, ίσως και το θέμα της ε, χρηματοδότησης της έρευνας ή της πρόθεσης της έρευνας για καλύτερα, καλύτερη ποιότητα στην ανάλυση των δεδομένων. Επίσης θέλουμε και έγκαιρη εξαγωγή των πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων. Θέλουμε λοιπόν αυτή την πρόταση για την ενιαία διαπαφή για την αναζήτηση, για να είναι εύκολη και η εξαγωγή των δεδομένων από τις βάσεις και των πληροφοριών. Επίσης, συμφωνούμε ότι θα πρέπει να εξηγήσουμε διεξοδικά ε, τα ωφέλη ενός ενιαίου αποθετηρίου, ενιαίου κεντρικού αρχείου, αλλά πρώτα θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο κεντρικό αρχείο και μετά να πείσουμε για τα ωφέλη του. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρμαχος ενός τέτοιου κεντρικού αποθετηρίου, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε πιο διεξοδικά αυτό το θέμα. Συμφωνώ επίσης ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να... το έργο μας για τα θύματα και η εφαρμογή των μέτρων στην σχετική οδηγία θα είναι το επόμενο βήμα και ελπίζω να έχουμε κάποια στιγμή την ευκαιρία για πιο εμβριθή συζήτηση για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και τις γενικές απειλές ε, τέτοιων εγκλημάτων. Επίσης, αυτή η κυβερνοαθεκτικότητα που είπατε, η κυβερνοπροσαρμοστικότητα, είναι ένα θέμα που θα συγκεκριμενοποιείται στο μέλλον. Στην, την Άνοιξη, για παράδειγμα, θα υποβάλουμε προτάσεις για την ανάπτυξη μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Αρμόδιος είναι ο Αντιπρόεδρος Άνσιπ για το θέμα αυτό και θα υποβάλει σχετικές προτάσεις. Θα περιλαμβάνουν και ένα ειδικό κεφάλαιο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ανθεκτικότητα στα κυβερνοεγκλήματα. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο παρόλο που το άφησα για το τέλος και ελπίζω να μην ξέχασα τίποτα. Ασφάλεια της αεροπορίας. Ξέρω ότι το συζητήσατε και εσείς επανελειμμένως. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έλαβαν κάποια μέτρα, το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης κάποια μέτρα, κάπως διαφορετικά όμως. Και είχαμε επαφές με τις Βρετανικές αρχές ε, για τις αποφάσεις αυτές. Και θα έχουν την ευκαιρία την επόμενη εβδομάδα σε μια συνάντηση των εμπειρογνώμων για την ασφάλεια της αεροπορίας στις αρχές της επόμενης εβδομάδας να παρουσιάσουν διεξοδικά στους εταίρους τους το σκεπτικό ε, για τη λήψη αυτών των μέτρων. Από ό,τι ξέρω δεν ε, προκύπτουν από συγκεκριμένε ε, πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, αλλά περισσότερο από αξιολόγηση των ικανοτήτων κάποιων ομάδων που συνδέονται με την Αλκάιντα και αξιολόγηση των αντιμέτρων που οφείλουν να λάβουν. Αυτά θα το συζητήσουν όμως την επόμενη εβδομάδα οι εμπειρογνώμονες για την ασφάλεια στην αεροπορία και θα ενημερωθείτε εν καιρό για την έκβαση αυτής της συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Η κυρία Γκρίσπεκ είχε θέσει ένα ε, ερώτημα. Φαντάζομαι όμως ε, απαντήθηκε και φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι θα διαβιβάσουν την απάντηση αυτή στην ίδια. Ευχαριστώ πολύ και πάλι που αλλάξατε κάποια από εσά τουλάχιστον το πρόγραμμά σας για να είστε σήμερα εδώ. Θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας ε, με και με, τα, με τους εκπροσώπους ε, των κρατών μελών τη Δευτέρα για την εφαρμογή. Ε, καλό θα ήταν να παρευρεθείτε και σε εκείνη τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Επίτροπε, εσάς και το επιτελείο σας για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα και προσβλέπουμε στη συνέχεια που θα δοθεί ε, στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ.

Um, Συνάδελφοι, αν είστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο τελευταίο θέμα της σας διάταξης, σας ευχαριστώ και πάλι που είστε εδώ. Είναι μαζί μας και ο Λουίτζι Σορέκα, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Μιλούμε για, την, ε, για τις εκθέσεις εφαρμογής του PNR στις 9 ε, Φεβρουαρίου 19 Φεβρουαρίου η Κομισιόν εξέδωσε τις εκθέσεις εφαρμογής για το TFTP, το πρόγραμμα παρακολούθησης χρηματοδότησης τρομοκρατίας και το PNR ε, και επειδή ο πλέον αρμόδιος είναι ο ε, κύριος Σορέκα ε, θα κάνει τις παρουσιάσεις για αυτά τα θέματα. Είναι διευθυντής για θέματα ασφάλειας στη Γενική Διεύθυνση HOME Έχουμε μαζί μας ε, και άλλον έναν εκπρόσωπο. Ε, μάλλον ήταν ε, σχεδιασμένο να είναι κάποιος άλλος εδώ, αλλά ε, δυστυχώς λόγω των επιθέσεων του, του, του Λονδίνου δεν κατέστη δυνατόν. Παρ' όλα αυτά θέλω να την ευχαριστήσω. Δεν θα, δεν θα έχουμε την ευκαιρία λόγω της συνταξιοδότησης να την ξαναδούμε. Θα ήθελα να της διαβιβάσετε τις καλύτερες ευχές μου. Ε, κύριε Σορέκα. Λουίτζι, ε, έχεις το λόγο για να μας παρουσιάσει αυτές τις δύο εκθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη μου χαρά θα διαβιβάσω τις ευχές, ε, τις ευχές σας στην Πελίντα Πάιξ που συνταξιοδοτείται τώρα μετά από μια πολύ μεγάλη και επιτυχημένη καριέρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάφορα τμήματα. Βεβαίω και θα το κάνω. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μου δίνετε την ευκαιρία σήμερα να ε, παρουσιάσω τα αποτελέσματα των ε, δύο εκθέσεων εφαρμογής για τις συμφωνίες PNR και TFTP. Θα τα κάνω διαδοχικά ε, δίνοντας σας πληροφορίες για την κάθε μία από τις δύο συμφωνίες και στη συνέχεια θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί φυσικά να είναι ένα ευαίσθητο θέμα στην Ευρώπη και γι' αυτόν τον λόγο το να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται όλε οι δεσμεύσει και υποχρεώσει ε, που κατοχυρώνονται στι διεθνεί συμφωνίε που έχουμε διαπραγματευτεί εκ μέρου της Ένωσης και που επιτρέπουν τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων των πολιτών μα, ε, εφαρμόζονται σωστά είναι ζωτική σημασία για να εξασφαλιστεί ε, η προστασία ε, ε, των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και ότι τίθενται σε επεξεργασία με σύνομο τρόπο. Οι, στις κοινέ μας συνεδριάσεις με τους Αμερικανούς συναδέλφους είχαμε ένα πολύ επικοδομητικό πνεύμα. το PNR από την πλευρά της Ευρωπαϊκής, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, η οποία ε, της ευρωπαϊκής πλευράς μάλλον που αποτελούνταν από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και από εκπρόσωπο της γαλλικής ε, αρχής προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ε, μας έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβουμε πώ ακριβώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά από τους Αμερικανούς αλλά και μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε με ποιον ακριβώς τρόπο στοχεύουν σε συγκεκριμένες πληροφορίε. Η αναθεώρηση της ε, συμφωνίας TFTP έγινε με, υπό την αιγίδα του Επιτρόπου Φίσερ και με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων της Eurojust. Όπως γνωρίζετε, η έκθεση που έχετε στα χέρια σας είναι μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι ΗΠΑ είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν και εκείνες τα δικά του σχόλια για τις ε, δύο εκθέσεις αυτές. Και αυτό μας ε, επέτρεψε βεβαίως να λάβουμε υπόψη και τη δική τους οπτική και θα σας πω όμως σε λίγο και ποια ήταν τα σχόλια που δεν λάβαμε υπόψη μας, γιατί δεν συμμεριζόμασταν τις ε, απόψεις αυτές. Το βασικό πόρισμα λοιπόν ε, είναι ότι η εφαρμογή έχει στεφθεί γενικά με επιτυχία, ε, είναι σταθερή η συμφωνία όσον αφορά τις, τα εχέγγυα και τις δικλείδες ασφαλείας και αυτές θεωρούμε ότι εφαρμόζονται σωστά από τις Αμερικανικές Αρχές. Να ξεκινήσουμε με, το, με την έκθεση για το PNR μπορώ να σας πω ότι το, το, συνολικά, το συνολικό πόρισμα της αναθεώρησης είναι ότι οι ΙΠΑ ε, εφαρμόζουν τη συμφωνία σύμφωνα με, τον, ε, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που κατοχυρένονται σε αυτή τη συμφωνία. Όλες οι συστάσεις ε, που είχαν εκδοθεί πριν από τη συμφωνία από το 2013 και έπειτα έχουν ε, ληφθεί υπόψη ή έχουν υλοποιηθεί εφαρμοστεί και θα σας πω σε ποιες περιπτώσεις ζητήσαμε εμείς από τις Αμερικανικές Αρχές να, κάνουν περισσότερα από όσα έκαναν. Οι Αμερικανικές Αρχές σέβονται λοιπόν τις ε, προχρεώσεις τους όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και θέτουν σε επεξεργασία τα δεδομένα με βάση ε, τις δεσμές και τις υποχρεώσεις τους. Ε, η έκθεση αυτή μάλιστα θα, θα τροφοδοτήσει και την κοινή αξιολόγηση ε, της συμφωνίας η οποία θα μας δώσει μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη εικόνα ε, για την συμφωνία PNR. Για τα βασικά πορίσματα, γιατί δεν θα σας τα παρουσιάσω όλα, θα σας παρουσιάσω μόνο τα κύρια, τα βασικά πορίσματα, θέλω να επισημάνω σε εσά αυτά που εμείς θεωρούμε ότι είναι άξια λόγου. Όπως γνωρίζετε, ως προς το πεδίο ισχύω, η Συμφωνία PNR αφορά πτήσεις μεταξύ Ένωσης και ίπα αλλά έχουμε ε, επαληθεύσει ε, με θετικό τρόπο ότι οι ίπα εφαρμόζουν τις ίδιες απαιτήσεις προστασίας ε, για το PNR είτε πρόκειται για πτήσεις που έχουν ξεκινήσει εντός είτε εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όσον αφορά τα ίδια τα δεδομένα, το Υπουργείο Συντερικών των ΗΠΑ εξακολουθεί να χρησιμοποιεί αυτό το φίλτρο των 19 στοιχείων και ε, σε συνεργασία μας με τους ομολόγους μας από, την, από τις ΙΠΑ, μας ε, ε, ε, υπόθηκε ότι δεν, οι τελωνιακές αρχές των ΙΠΑ δεν έχουν παραβιάσει τις υποχρεώσεις τους. Όσον αφορά το άρθρο 5 και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και εδώ οι αρχές έχουν εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο εργαλείο που το αποκαλούν CBT Custom Control Border, Border Control προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι το PNR ε, είναι προστατευμένο και ότι μόνο άτομα εξουσιοδοτημένα έχουν πρόσβαση σε αυτό. Δεν έχουμε ε, εντοπίσει περιστατικά που να αφορούν ε, παραβίαση προσωπικών δεδομένων Ευρωπαίου πολίτη για την περίοδο μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης αναθεώρησης. Έχουμε επαληθεύσει τη διαγραφή και την ανωνυμοποίηση ε, δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 και το Υπουργείο Ιστορικών των ΗΠΑ μας είπε ότι δεν, ε, έχουν ποτέ αποκτήσει, δεν είχαν ποτέ πρόσβαση, ε, δεν έχουν ποτέ προσπελάσει ευαίσθητα δεδομένα. Υπάρχει ένα θέμα διαφάνειας όσον αφορά την συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Ευρωπαίων πολιτών. Εδώ πράγματι έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εύρος πληροφοριών ε, που είναι δημόσια ε, διαθέσιμος στις, ε, στο διαδίκτυο και έχουμε ζητήσει από τους Αμερικανούς ομολόγους μας να τηρήσουν οπωσδήποτε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία για το PNR. Κανένας πάντως επιβάτης δεν έχει μέχρι στιγμής ζητήσει τη διαγραφή ή την διόρθωση των στοιχείων του. Τέλος, Όσον αφορά την, ε, την πράξη για τα ένδικα μέσα, για την νομική προσφυγή που τέθηκε σε εφαρμογή το 2015, πράγμα, έχει και αυτή τεθεί σε εφαρμογή ε, όσον αφορά το PNR. Και αυτό είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη που θεωρώ ότι και το Κοινοβούλιο μπορεί να αναγνωρίσει. Ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους χρειάζεται πιο πολύ δουλειά. Ας ε, επικεντρώσουμε λοιπόν σε αυτά τα ζητήματα. Η ομάδα της Ένωσης έκανε δέκα συστάσεις. Πρώτον, ε, προτείνουμε τη βελτίωση της στήρισης αρχείων, κάτι που θα βοηθήσει να, να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της, ε, συμφωνίας. Ε, Ιδίω όταν διαβιβάζονται πληροφορίες των PNR σε άλλες, ε, σε τρίτες υπηρεσίες. Επίσης, προτείναμε το DHS, ε, το Υπουργείο Εσωτερικών, τον είπα να, να διερευνήσει για ποιο λόγο δεδομένα της, του PNR έχουν συσχετιστεί με άσχετες υποθέσεις. Ε, ξέρουμε ότι έχει γίνει έργο στον τομέα αυτόν ε, ε, από την τελευταία αναθεώρηση και έπειτα, άρα νομίζουμε ότι αυτή η σύσταση έχει πραγματικά υλοποιηθεί. Όσον αφορά την πρόσβαση στο PNR, είναι ένα ζήτημα που επίσης έθεσε η δική μα ομάδα. Αυτό ήταν πρόβλημα που είχε διαπιστωθεί το 2013. Δυστυχώς εξακολουθεί να είναι πρόβλημα, ε, ήταν, ε, εξακολουθούσε να είναι πρόβλημα και το 2015. 2.000 άτομα έχουν ε, δικαιώματα πρόσβασης στο PNR. Μας υπόθηκε ότι αυτό οφείλεται σε σκοπούς εποπτείας, εκπαιδευτικού σκοπού. Ζητήσαμε διευκρινήσει από του Αμερικανού και θα εξετάσουμε τα ζητήματα αυτά κατά τη διάρκεια της ε, επικείμενης ε, κοινή αξιολόγησης. Η κοινή αξιολόγηση λοιπόν είναι κάτι διαφορετικό από την κοινή έκθεση. Την κοινή αναθεώρηση. Ε, συγγνώμη. αφορά την... είναι μια δέσμευση που προβλέπεται στην ίδια συμφωνία, ενώ η, η κοινή αξιολόγηση έχει ευρύτερο σκοπό. Ε, έχει σκοπό να εξετάσει αν ε, ικανοποιείται, αν, αν ε, επιτυχάνεται ο στόχος, της, ο βασικός στόχος της συμφωνίας και αν εξακολουθεί να είναι κατάλληλο εργαλείο. Αυτό ήταν και αίτημα του Κοινοβουλίου. Ακόμη και αν η κοινή αξιολόγηση έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί το 2016, θέλαμε να περιμένουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το σχέδιο συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά προκειμένου να συγκρίνουμε την κοινή αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια που θα μας έδινε τότε το, δικαστήριο προκειμένου να έχουμε μια συνοχή και συνέπεια ε, στην κοινή αξιολόγησή μας και να μην δημιουργηθούν προβλήματα και το ξεκαθαρίσαμε αυτό και στους Αμερικανούς ομολόγους μας. Κλοντ, αν μου επιτρέπεις τώρα, θα ήθελα να περάσω και στην συμφωνία TFTP agreement as well, we... Η συμφωνία βαίνει καλώς. Πρέπει να πούμε ότι εφαρμόστηκε καταλήλως και τα απορίσματα της προηγούμενης κοινή αναθεώρησης ε, τα συζητούμε με τις Αμερικανικές αρχές. Η συμφωνία TFTP ε, ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο τα τελευταία δύο χρόνια ε, για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως την Ευρωπόλ αλλά και για τις εθνικές ε, αρχές ε, για να μπορέσουν να κάνουν έρευνες ε, για τις επιθέσεις οι οποίες, επιθέσεις οι οποίες έγιναν στην Ευρώπη. Στο παρελθόν φαντάζομαι ότι λάβατε και ενημέρωση. Τα διάφορα στοιχεία τα οποία έδωσε η TFTP στις αρχές επιβολής του νόμου αποτελούν μαρτυρία αυτής της καλής εφαρμογής. Όσον αφορά τα πορίσματα, η έκθεση επιβεβαίωσε ότι οι δύο μηχανισμοί ελέγχου που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο ένας της Ευρωπόλ και ο άλλος ε, ε, των Ευρωπαίων ελεγκτών που ε, όρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν αποτελεσματικά, η Ευρωπόλ ε, τηρεί τα καθήκοντά τη και ο έλεγκτοχος και η εποπτεία λειτουργεί αποτελεσματικά και ε, αποδοτικά. κάτι το οποίο θα ήθελα να σας επισημαίνω είναι ότι ο χρόνος διατήρησης, ο οποίος βάσει της συμφωνίας είναι το πολύ πέντε χρόνια, γίνεται σεβαστός και το επαληθεύσαμε αυτό, μας δόθηκε ευκαιρία να το επαληθεύσουμε. Σε γενικές γραμμές λοιπόν είναι ικανοποιητική η έκθεση και ζητήσαμε από τους Αμερικανούς να κάνουν κάποια περισσότερα ε, διότι τους ζητήσαμε να έρθουν ε, περαιτέρω σε επαφή με τα κράτη-μέλη μέσω της Ευρωπόλ ώστε να χρησιμοποιείται ακόμα πιο εκτεταμένα ε, το σύνολο αυτών των εργαλείων, τα οποία όπως είπαμε ήταν πάρα πολύ σημαντικά ε, στις πιο πρόσφατες επιθέσεις και μπορώ να πω και στην χθεσινή επίθεση στο Λονδίνο. Οι έλεγχοι του TFTP ε, που ζητήθηκαν από τα κράτη-μέλη που ενεπλάκησαν ε, διαβιβάστηκαν στις αγγλικές αρχές. Θα σταματήσω εδώ κύριε Πρόεδρε, εάν συμφωνείτε. Νομίζω ότι μίλησα 17 λεπτά και πολύ ευχαρίστως θα απαντήσω και στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ Λουίτζι για αυτή την ε, συνολική ε, αναφορά που μας έκανες. Ε, οι συνάδελφοι είναι εδώ και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παραμείνατε. Συγγνώμη που έχουμε τόσα πολλά πράγματα στην ημερήσια διάταξη αυτή την εβδομάδα και το εκτιμώ το γεγονός ότι παραμείνατε. Ποιος θέλει να πάρει πρώτος το λόγο. Η Μπίρκη είχε ζητήσει το λόγο, η Σόφη, η Μόνικα θα μιλήσει. Τι κάνω, κουράζομαι και σας ρωτάω αν θέλετε να μιλήσετε. Τι κάνω, τα έχω χάσει. Ζητώ συγγνώμη, ήταν πολύ δύσκολη η κουραστική εβδομάδα. Μπίργκιτ, θέλει να μιλήσει. Ευχαριστούμε πολύ για την έκθεση αυτή. Χαίρομαι που ακούω ότι τα θέματα της εφαρμογής και τα καθήκοντα σε γενικές γραμμές φαίνεται να πηγαίνουν καλώς. Ε, ε, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, εντάξει, κάποιες εκκρεμότητες και από ό,τι κατάλαβα η ευρύτερη εικόνα που θα γίνει μέσω της αξιολόγησης δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω κάποιες ερωτήσεις, ε, αν μπορείτε, διότι αν δεν τα είχατε στην αξιολόγηση, ίσως θα μπορούσατε να τα λάβετε υπόψη για την επόμενη αξιολόγηση. Ένα από τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι ότι εντάξει, τα έχουμε εφαρμόσει λίγο πολύ, ε, λειτουργούν. Το θέμα είναι ε, πόσο σημαντικά είναι αυτά τα μέτρα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ε, πριν από κάποιο καιρό είχα δει κάποια στατιστικά στοιχεία για το πόσες ε, θετικές ε, απαντήσεις είχαμε για υπηκόους κρατών μελών που εξέτασαν τα στοιχεία PNR, αλλά ποτέ δεν είδα στατιστικά στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη, τα οποία μπορεί να οδήγησαν σε έρευνα ή ε, αποτέλεσαν και αντικείμενο ε, έρευνας που οδήγησε σε πληροφορίες ε, για το οργανωμένο έγκλημα ή την τρομοκρατία. Μήπως έχετε κάποια γενικότερα σχόλια να κάνετε για το τι ε, ακριβώς έχει πετύχει το PNR. Όσον αφορά την TFTP, υπάρχει αυτή η γενικότερη άποψη ότι πάντα καλό είναι, αν θέλει κάποιο να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα, ε, πρέπει να ακολουθήσει το χρήμα. Αυτή είναι η γενικότερη άποψη που επικρατεί. Και πάλι όμως ε, το θέμα είναι, έχει αποτέλεσμα αυτό και αν θέλουμε να τα δούμε ευρύτερα, όχι μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείε Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ε, γενικότερα στο διεθνέ οργανωμένο έγκλημα και στην τρομοκρατία διότι ε, πολύ συχνά και οι δύο τομείς είναι αλληλένδετοι. Τα μέτρα αυτά και τα δύο μας δίνουν περισσότερες γνώσεις για το τι συμβαίνει, ιδιαίτερα για την DFTP Πρόκειται για εργαλείο το οποίο βοηθά να σταματήσει τουλάχιστον κάποιες μορφές χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ε, το 100% δεν θα το καταφέρουμε ποτέ, αυτό είναι σαφές, αλλά καταφέραμε τα τελευταία χρόνια να έχουμε κάποιες πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να σταματήσουμε κάποιες μορφές χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Θα ήταν χρήσιμο αυτό. Ευχαριστώ η Μόνικα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τρία ερωτήματα θέλω να θέσω. Πρώτον, υπάρχουν κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν ήδη το PNR και έχουν συλλέξει και κάποια, ε, κάποιες εμπειρίες. Σε ποιο βαθμό λειτουργεί εύρυθμα αυτή η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών ή να το πω αλλιώς ενδεχομένως ποια προβλήματα έχουν εμφανιστεί ε, γιατί κάτι τέτοιο θα μας βοηθούσε ενδεχομένως να προβλέψουμε και τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν ε, όταν όλα τα κράτη-μέλη ε, εφαρμόσουν το PNR. Γιατί σε τελική ανάλυση χρειάζεται, αυτό που στόχος είναι να δημιουργηθεί μια κοινή βάση δεδομένων και μια αποτελεσματική χρήση των δεδομένων αυτών. Χθες στη διάσκεψη ε, της Ευρωπόλ, ο καθηγητής Νόιμαν ε, ανέφερε ότι πρόβλημα ε, είναι και οι μικροχρηματοδοτήσεις και όχι μόνο τα μεγάλα χρηματικά ποσά που κατευθύνονται στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Είναι τα μικρά μικρά ποσά δηλαδή που συλλέγονται από διάφορους υποστηρικτές. Υπάρχουν ε, δεδομένα για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τέτοιου είδους ε, στοιχεία ή πληροφορίες για την ταυτοποίηση μικροεγκληματιών ενδεχομένως ε, γιατί βλέπουμε και από τα χθεσινά γεγονότα στο Λονδίνο ότι πολλές φορές δεν χρειάζεται καν να έχει κάποιος φοβερά μέσα χρηματικά στα, στα χέρια του. Αρκεί και ένα μαχαίρι πολλές φορές. Για το TFTP θέλω επίσης να ρωτήσω κάτι. Ε, συμμετέχουν βεβαίως και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ε, μαζί με ε, ε Αμερικανούς. Πότε πιστεύετε ότι θα έχουμε εμείς κάποια στιγμή την ικανότητα να συστήσουμε ένα δικό μας ευρωπαϊκό TFTP αντί να διαβιβάζουμε διαρκώς τις πληροφορίες τους Αμερικανούς και στη συνέχεια εκείνοι να μας ξαναστέλουν πίσω τα δεδομένα επεξεργασμένα. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερα αν μπορούσαμε ε, να επεξεργαζόμαστε εμείς τα δεδομένα αυτά και στη συνέχεια σε, αυτό, σε ισότιμη βάση να τις ανταλλάσσουμε τις πληροφορίες αυτές με τις ΕΙΠΑ. Ευχαριστώ πολύ, Σόφι Ιντβελτ. Ευχαριστώ. Και εγώ συνεχίζω το τελευταίο σχόλιο. Όταν έγιναν οι δύο συμφωνίες, FTP και PNR, Είχαμε ρωτήσει γιατί να μην κάνουμε εμεί την αναζήτηση και να δώσουμε κατευθείαν στου Αμερικανού τα στοιχεία που χρειάζονταν και μα είπαν ότι ήταν οικονομικό το θέμα. Τελικά αυτό γινόταν γιατί είχαμε, ε, ετοιμάζαμε τότε τα δικά μας στήματα που ήταν ακόμη πιο αυστηρά. Εγώ δεν φανταζόμουν τέτοιε εξελίξει. Σε ό,τι αφορά την πράξη για, την, για τα ένδικα μέσα, αυτό ισχύει και για το PNR είναι αρκετή FTP ή μήπως σας παρεξήγησα. Γιατί υπάρχει εδώ μία ζώνη του λυκόφωτος ό,τι αφορά τις πληροφορίες που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αρχικά έχει αναγνωρίσει ότι το PNR και το TFTP είναι συστήματα που ε, εξαιρούνται από τον ε, νόμο για την ε, ιδιωτικότητα, κάτι όμως που δεν συμπίπτει με τον νόμο για τα άδικα μέσα. Φαίνεται ε, εσκεμένα να μπερδεύει τα δύο, τις δύο νομοθετικές πράξεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. θα πρέπει να διευκρινιστεί αυτό γιατί είναι σημαντικό ζήτημα. Ε, θα το στείλω και γραπτό με επιστολή, αλλά μπορείτε να μας το εξηγήσετε και τώρα. Επιβεβαιώστε δηλαδή ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν αποφασίσει ακόμη ή δεν έχουν ακυρώσει την εξαίρεση του PNR και του TFTP από την νομοθετική πράξη για την ιδιωτικότητα. Και συμφωνείτε ότι αν κάτι τέτοιο ισχύει η Γενική Συμφωνία δεν ισχύει και η νομοθετική πράξη για τα 11 μέσα ε, δεν έχει καμία σχέση με την πράξη για την ιδιωτικότητα. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Γιούντι Σαρσεντίνη. Ευχαριστώ. Κατάλαβα καλά ότι ακόμη ούτε ένας επιβάτη δεν ζήτησε τα στοιχεία του για το PNR ή μήπω δεν σας κατάλαβα καλά, γιατί αν κατάλαβα καλά, πού πιστεύετε ότι οφείλεται κάτι τέτοιο, ότι κανείς δεν ζήτησε να δει τα στοιχεία του ή να ζητήσει αφαίρεση το στοιχείο του από το σύστημα. Μήπως ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι τα στοιχεία του είναι μέσα σε ένα σύστημα. Είπατε ότι περιμένετε ακόμη ε, την απόφαση του ΔΕΚ για το PNR με τον Καναδά. Και εμείς περιμένουμε με περιέργεια αυτή την ομολογία. Πάντως φαίνεται ότι ο Γενικός εισαγγελέα είναι πολύ σχολαστικός ε, και δεν ξέρω τι θα σημάνει μια τέτοια δικαστική απόφαση στις ε, διαπραγματεύσεις με την Κορέα, το Μεξικό ή την Ιαπωνία γιατί ακόμη συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τις χώρες αυτές. Σε ό,τι αφορά το TFTP, ειλικρινά σας λέω ότι είναι η πρώτη φορά που μας λέει ένας υπάλληλο, ίσως ε, κατά λάθο, μας είπατε ότι από τη χθεσινή ε, τρομοκρατική επίθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, δεν είχε ζητηθεί κάτι τέτοιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι η πρώτη φορά που κάποιο ε, ε, υψηλά ιστάμενο μας λέει για το πώς χρησιμοποιούνται τέτοια στοιχεία. Μακάρι να μιμηθούν και άλλοι το παράδειγμά σας, έστω και αν έγινε από παραδρομή. Γιατί ακόμη περιμένουμε ε, μία έμπρακτη απόδειξη της χρήσης του, του συστήματος TFTP. Επίσης έγινε συζήτηση για ένα ευρωπαϊκό TFTS σε ποια φάση της συζήτησης είμαστε. Δεν είμαι και πολύ θυσιώδης για το θέμα αυτό. Αλλά αν έτσι ξεπεράσουμε τα θέματα προστασία δεδομένων που έχουμε με τις ΗΠΑ, ίσως τάξει το κόπο να το διερευνήσουμε περαιτέρω. Ευχαριστώ. Η Χέλγα Στίβενς έχει τώρα το λόγο και δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλος που θα ακολουθήσει. Όχι, η τελευταία είναι η Χέλγα Στίβενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίασή του για το TFTP και το PNR. Χρήσιμες πληροφορίες και θα πρέπει να συνεχίσουμε την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών, φυσικά αναζητώντας και βρίσκοντας τη σωστή ισορροπία μεταξύ της χωρίς πληροφοριών για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας της ιδιωτικότητας γιατί είναι πολύ λεπτή αυτή η ισορροπία φορές. Από ό,τι φαίνεται προς το παρόν το σύστημα περιορίζεται στους ε, επιβάτες των αεροπορικών εταιριών. Προτάθηκε όμως ε, να επεκταθεί και στις ε, διεθνείς σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές με πούλμαν. Ποια είναι η γνώμη σας Υπάρχουν καταρχήν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να έχουν εγκρίνει αυτό το διάβημα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογή ή θα περιοριστούμε μόνο στους, α, στις αερομεταφορές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Σορέκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και όλα τα μέλη της ε, Επιτροπής για τα ερωτήματα που θέσατε. Θα ξεκινήσω, θα απαντήσω με τη σειρά που τέθηκαν. Κάποια μάλιστα ήταν και παρόμοια, εν μέρη τουλάχιστον. Όσον αφορά τα δεδομένα και τα αποτελέσματα, τα hits που χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη ε, στο PNR, αλλά και στο TFTP, με, με άλλο τρόπο, συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την, την, της, τον αριθμό των ε, επικλήσεων της, της συμφωνίας. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι όταν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το PNR, τα κράτη-μέλη θα είναι πλέον πιο πολύ εκπαιδευμένα ε, και πιο εξοικειωμένα με το να αξιοποιούν τις πληροφορίες που θα απορρέουν από τις διεθνείς μας συμφωνίες. Χρειάζεται χρόνος μέχρι να ριζώσει ένα τέτοιο σύστημα, αλλά όταν αυτό γίνει ε, είναι βέβαιο ότι και τα δεδομένα που θα απορρέουν από τις συμφωνίες μας θα είναι πιο ε, χρήσιμα. Στο TFTP τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Ε, λόγω και, του ρόλου που διαδραβάτησε η Ευρωπόλ στο TFTP. Η Ευρωπόλ έχει το ρόλο φιλτραρίσματος των δεδομένων και γι' αυτό έχει και το δικαίωμα ε, να αναλάβει την πρωτοβουλία, να επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ προκειμένου να, συγκεντρώσει δεδομένα κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους και στη συνέχεια να επαναπροωθήσει αυτά τα δεδομένα στο εν λόγω κράτος μέλους. Ε, μπορώ βεβαίως να σας τα στείλω αυτά και επισήμως. για το αν το TFTP ε, κατάφερε να σταματήσει κάποια μορφή χρηματοδότησης ε, της τρομοκρατίας, κάτι που συνδέεται και με αυτό που είπε η κυρία Χόλμαϊρ για την μικροχρηματοδότηση. Είναι αλήθεια ότι, ότι στις τελευταίες τρομοκρατικές επιθέσεις οι τρομοκράτες δεν χρησιμοποίησαν τεράστια ποσά. Ε, είχαν λάβει ε, βεβαίως ε, σημαντικά χρήματα για την, ε, για την εκπαίδευσή τους και για να διοργανώσουν τις, για να οργανώσουν τις επιθέσεις, αλλά για την ίδια την, τη στιγμή, την ημέρα της επίθεσης δεν χρειάστηκαν πολλά χρήματα. Αυτό είναι αλήθεια και συνάδει με μια ανάλυση της Κομισιόν του 2013, η οποία έλεγε ότι το TFTP ε, δεν ήταν κατάλληλο ε, για πολλούς λόγους, για λόγους κόστους για παράδειγμα ή για λόγους ε, αποτελεσματικότητας. Όμως η κατάσταση ως προς την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει. Έχετε ακούσει πολύ συχνά ότι πλέον έχουμε ε, εγχώρια τρομοκρατία, ριζοσπαστικοποιημένους ανθρώπους και πλέον ε, ε, έχουμε το πρόβλημα αυτό εντός της Ευρώπης και γι' αυτόν τον λόγο η Κομισιόν ξεκίνησε μια αξιολόγηση στο πλαίσιο του σκεπτικού να δημιουργηθεί ένα EUTFTS στην έκθεση προόδου του Επιτρόπου King στις αρχές του χρόνου αναφέρεται ότι έχει ξεκινήσει το σχετικό έργο και ξέρετε ότι ε, προετοιμάζεται και μια μελέτη επιπτώσεων προκειμένου να ε, στραφούμε σε εσάς ε, προς το τέλος του έτους με συγκεκριμένη ή και χωρίς συγκεκριμένη πρόταση για ένα ευρωπαϊκό TFTS που θα καλύπτει εκείνες τις, εκείνους τους τομείς που δεν καλύπτονται από το TFTP. Με άλλα λόγια θα έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα και θα αποτελεί ε, στην πραγματικότητα ένα ευρωπαϊκό TFTF. Όσον αφορά τα ένδικα μέσα, και συγγνώμη αν δεν τα εξήγησα σωστό, ε, αυτό που είπα είναι ότι η θέση σε ισχύ της ε, εν λόγω πράξης το 15 μετά την ε, αξιολόγηση ήταν μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη ε, ακόμη και αν η συμφωνία, ε, η Γενική Συμφωνία δεν τέθηκε αμέσως σε εφαρμογή. Θα μας βοηθήσει όμως τις, από εδώ και πέρα αξιολογήσεις μας, οι οποίες θα γίνουν στο δεύτερο εξάμεινο του 2017, προκειμένου να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα και των ασφαλιστικών δικλείδων του PNR υπό το πρίσμα και αυτής της Τη εφαρμογή αυτής τη ε, νομοθετική πράξη. Όσον αφορά την κυρία Σαρτζεντίνη, κανείς πράγματι δεν έχει ε, ζητήσει την επικύρωση των ε, δεδομένων που έχουν διαβιβαστεί. Αυτό μας έχει, αυτό γνωρίζουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα σε διάφορες ιστοσελίδες των τελωνίων και από αυτή την άποψη πράγματι υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια ε, που δίνουν την, τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν δεδομένα ε, επιβατών και αυτό πρέπει να το δούμε. Όσον αφορά την, τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, μία είναι η ανοιχτή διαπραγμάτευση, που είναι η διαπραγμάτευση με το Μεξικό, για την οποία η Κομισιόν έχει λάβει εντολή το 2015. Φυσικά, Έχουν ανασταλεί οι διαπραγματεύσει έως ότου εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου. Φυσικά υπάρχουν και κάποιες συζητήσεις με την Κορέα και την Ιαπωνία, αλλά είναι τελείω άτυπε αυτές οι συζητήσεις. Έχουμε ξε, ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να γίνει διαπραγμάτευση προτού εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου και πρωτού ε, προτού δημοσιοποιηθεί και η, εκτίμηση του δικαστηρίου. Όσον αφορά τις ε, διεθνείς μεταφορές, ξέρετε ότι ε, η συμφωνία PNR και ε, ο κανονισμός δεν προβλέπουν την ε, κάλυψη άλλων τρόπων μεταφορέας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια αξιολόγηση για το αν κάτι τέτοιο θα ήταν χρήσιμο. Ε, πάντως η Κομισιόν αυτή τη στιγμή μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν, δεν έχει αναλάβει κάποια δράση ούτε επιτυλεί κάποιο έργο ε, ως προς ε, μια τέτοια πιθανή νομοθετική ρύθμιση. Θα αξιολογήσουμε, συλλέγουμε τις πληροφορίες και θα αξιολογήσουμε ε, ένα τέτοιο ενδεχόμενο με βάση την αναλογικότητά του. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Λουιτζή. Πολύ σύντομα η Σόφη Ινεντβέλτ θέλει μια επερώτηση. Θα ήθελα κάποιες εξηγήσεις γραπτός για την κατάσταση τώρα, διότι για τη συμφωνία, τη συνολική, θα αφορά και το PNR και το TFTP. Νομίζω ότι εσείς είπατε ακριβώς το αντίθετο. Το θέμα είναι ότι τμήμα του όλου οικοδομήματος, η συμφωνία συνολική, η, τα ενδικά μέσα κλπ. ήταν η ανάκληση των εξαιρέσεων στην πράξη για την ιδιωτικότητα για το PNR και το FTP. Βέβαια, εγώ δεν θα πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό ποτέ, δεν θα το κάνουν οι Αμερικανοί, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε γραπτός μάλιστα ότι αυτό θα γίνει. Κάθε φορά που προσπαθώ λοιπόν να το θίξω σε συζήτηση, σε επιστολές, σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, όλα γίνονται πολύ αόριστα. Διότι φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρει καν τι κάνει. Πραγματικά λοιπόν θα το εκτιμούσα, θα ήθελα να μου δώσετε γραπτός μία απάντηση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι διάφορε απαντήσει από τι διάφορε γενικέ διευθύνσει και διάφορε επιτρόπε. Μία απάντηση, μία εξήγηση. Πού βρισκόμαστε, συνολική συμφωνία ένδικα μέσα ανάκληση των εξαιρέσεων για την ε, νομοθεσία για την ιδιωτικότητα. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Και η Birgit πολύ σύντομα και μετά θα ολοκληρώσουμε. Πολύ σύντομα ζητώ συγγνώμη εάν δεν εκφράστηκα σωστά όσον αφορά τα θετικά αποτελέσματα στο PNR. Η ερώτησή μου ήταν ότι ναι, γνωρίζω ότι πότε πότε σε μια αξιολόγηση μας δίνουν την πληροφορία ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε μας είπαν ότι δόθηκαν κάποιες πληροφορίες στα κράτη-μέλη για πιθανές ε, ποινικέ διαδικασίες, άρα είχαμε κάποιες θετικές απαντήσεις, κάποια χιτ. Ε, αυτό που δεν ξέρω είναι τι τις έκαναν αυτές τις πληροφορίες στα κράτη-μέλη. Έκαναν κάτι, όντως, ε, και κατά πόσον έγινε και ποινική έρευνα στη συνέχεια ή αν υπήρξε κάποια δικαστική απόφαση. Είμαι βέβαιη ότι δεν άκουσα τίποτα για κοινοβούλια κρατών μελών που παρακολούθησαν ε, τις εξελίξεις. Το θέμα είναι κατά πόσον είναι αποτελεσματικά λοιπόν, τα χρησιμοποιούμε, ελέγχουμε αν υπάρχει κάτι όταν οι Ηνωμένε Πολιτείες μας δίνουν πληροφορίες ή απλώς ε, τα πετάμε στον κάλαθο των αχρήστων και δεν τα κοιτάει κανείς. Η κυρία Βερζιά, πολύ σύντομα παρακαλώ, πραγματικά πολύ σύντομα. Δεν ε, θα καταχρωστώ το χρόνο μιλίας κύριε Πρόεδρε, μην ανησυχείς. Η απάντηση που μόλις δώσετε στην κυρία Σαρχεντίνη με εντυπωσίασε. Άκουσα την... Είχα την ίδια αντίδραση μαζί της όταν σας άκουσα. Είπατε ότι δεν υπήρχε αίτημα πρόσβαση στα δεδομένα και αίτημα διόρθωσης των δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι όλα πάνε καλά ή μήπως θα έπρεπε να αναρωτηθούμε μήπως υπάρχει πρόβλημα διότι είναι μία από τις πολύ μεγάλες ανησυχίες μας όταν θα επίθετο το θέμα της εφαρμογής της συμφωνίας, της πληροφορίας και την ίδια τη δυνατότητα που έχουν οι πολίτες να έχουν πρόσβαση, να ξέρουν πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση και να ζητήσουν και διόρθωση. Και τι εγγύησεις έχετε επί του θέματος. Ναι, στην κυρία Ενέτβελτ. Βεβαίως. Ε, από ό,τι κατάλαβα, μας γράφετε επιστολές και σίγουρα θα πάρετε απάντηση από ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνολικά. Διότι όπως μας είπατε και δικαίως, πρόκειται για σύνθετο ζήτημα το οποίο ε, αφορά αρκετά τμήματα. Άρα, σαφέστατα και θα λάβετε απάντηση. Στην κυρία Ζίπελ. Παρακολούθηση δεν έχουμε πληροφορίες για το κατά πόσον τα κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν και πώς χρησιμοποίησαν αυτές τις πληροφορίες. Νομίζω ότι όλο και περισσότερο κατά την εφαρμογή της οδηγίας ε, PNR η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σαφέστατα διαδραματίζει ρόλο επ' αυτού, θα μπορέσει να απαντήσει στην ερώτησή της σας. Και τέλος, ε, Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι DHS, ε, το τμήμα εσωτερικής ασφαλείας των ΗΠΑ, δίνει αρκετές πληροφορίες στους επιβάτες μέσω των ε, πληροφορών που διατίθεται στο αεροδρόμιο, μέσω των πληροφορών που διατίθεται στην ιστοσελίδα προς όλους τους επιβάτες. Το έχουμε ζητήσει ε, επισήμως κατά πόσον υπάρχει σχετική τεκμηρίωση και μας είπαν ότι κανένας επιβάτης στην πραγματικότητα δεν έχει χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα μέσα, τα οποία όμως είναι διαθέσιμα. Ευχαριστώ Λουίτζι. Θα σταματήσουμε εδώ. Να ευχαριστήσω θερμά τον Λουίτζι και όλους εσάς. Ήταν μια μακρά δύσκολη εβδομάδα για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, και εσάς και το προσωπικό. Γιατί εσείς δεν έχετε επιλογή, εδώ πρέπει να είστε. Ε, ε, είστε σαν τη βασίλισσα, δεν μπορείτε να απαντήσετε, πρέπει να κάθεστε στη θέση σας. Ήταν λοιπόν πολύ έντονη η εβδομάδα για όλους. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν που ήσασταν εδώ. Ε, κάτι αντίστοιχο θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα και η ζωή συνεχίζεται. Καλό Σαββατοκύριακο και σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας.